Um, uh, Μπορούμε να αρχίσουμε παρότι είναι ακόμη απόντες πάρα πολύ, αλλά ε, έχουμε καθυστερήσει ήδη αρκετά και είναι φορτωμένη η μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να αρχίσω με το πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυρία Ουκατσιεύσκα έχει υποβάλει ένα αίτημα και θα ήθελα τη δική σας έγκριση να μετατε... Στο σημείο 8, επειδή είναι σκιώδης για το ΕΛΚ, θέλει να μεταφερθεί και δεν θα μπορέσει να μιλήσει ε, αν παραμείνω σε έχει διάταξη και θέλει, ζητάει να μεταφερθεί και να μπει μετά το σημείο 5, αν συμφωνείτε. αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνεται. Η μερίσια διάταξη αναμεταδίδεται ως συνήθως η συνεδρίαση. Να το λάβετε υπόψη παρακαλώ. Επίσης είναι δεικτικό το χρονοδιάγραμμα, μπορεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ε, να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κάθε μεμονωμένο σημείο. Ωραία, τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών συνεδρίαση τη προηγούμενη ε, συνεδρίαση, μάλλον στι 14 Οκτωβρίου. Έχουν μοιραστεί τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα με το πέρα τη συνεδρία, αν δεν προβάλλεται στάση κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση. Και περνώ στο σημείο 3. Ανακοινώσει ε, τη Προέδρου. Ο Λαμπέρ θέλει να μιλήσει, αλλά μήπως να κάνω και εγώ τις ανακοινώσεις πρώτα που έχω, όπως το έχω σχεδιάσει, ωραία. Προχθές ε, και χθες, ε, Δευτέρα και Τρίτη, ε, ήμουν στο Βίλνιους. Μας είχε προσκαλέσει για δύο εκδηλώσεις η Προεδρία τη Δευτέρα. Για πρώτη φορά συζητήσαμε στη Βουλή με τους Προέδρους δύο επιτροπών. Εκπροσωπήθηκαν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιβάλλοντας και το θέμα ήταν η μακροπεριφαρία σε στρατηγικές, όχι μόνο στην περιοχή της Βαλτικής, αλλά γενικότερα. Εγκρίθηκαν ε, και συμπεράσματα σε συνεδρία, τα οποία θα μοιράσουμε σε όλους σας. Εν γέννη, ομολόγω, α, ήταν και ο Επίτροπος Χάντεχη, εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε διάφορες ε, επιμέρους συνόδους της διάσκεψης. Προετοιμάζοντας τα συμπεράσματα, Προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε κάποιες συστάσεις προς την μελλοντική Προεδρία για κοινέ δραστηριότητες με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών που είναι της αρμοδιότητάς μας για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό φυσικά θα είναι συνάρτηση της πολιτικής ε, των μελλοντικών, ε, της μελλοντικής προεδρίας. Εχθές έγινε άτυπο συμβούλιο. Οι υπουργοί ε, περιφερειακής πολιτικής και ε, αρμόδιοι για θέματα συνοχής ε, συσκέφθηκαν. Προηγούμενο συμβούλιο έγινε επί Κυπριακής Προεδρίας εχθές συζητήθηκαν οι προκλήσεις ε, κατά την εφαρμογή της πολιτικής. Ο Επίτροπος Χαν παρευρέθη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διάφορες περιφερειακές ε, οργανώσεις εκπροσωπήθηκαν επίσης. Ε, αυτές οι, οργαν... η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επίσης εκπροσωπήθηκε. Νομίζω ότι ο στόχος ήταν ε, να διαπιστωθεί ποια πρόοδος έχει σημειωθεί στα διάφορα κράτη-μέλη για την ε, προετοιμασία της ε, μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής. Δεν έχουμε ακόμη τα συμπεράσματα στη διάθεσή μας με το που καταφθάσουν ο Μιγγέλ ε, θα σας μοιράσει τα συμπεράσματα, θα δείτε ποια ήταν τα πορίσματα της ε, ε, συνεδρίασης. Νομίζω ότι όλοι τόνισαν πόσο δύσκολες δύσκολες ήταν οι εργασίες και χαίρονται που επι, επιτέλους θεσπίστηκε το, το πλαίσιο κατόπιν αιτήματός μας για την όλη διαδικασία των κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων ε, εκφράσαμε την ε, βούλησή μας ε, με εμπιστοσύνη να συνεργαστούμε και τελικά εγκρίναμε το σχέδιο και πριν τα Χριστούγεννα θα συγκληθεί και η ομάδα εργασίας για την πολιτική συνοχής για να ε, τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το θεματολόγιο για την εφαρμογή της διαδικασίας κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και ε, πώς ακριβώς ε, θα διαμορφωθεί η μελλοντική συνεργασία μας. Αρχίσαμε με τη Λιθουανική Προεδρία, αλλά το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στην Ελληνική Προεδρία. Τι άλλο να πω γι' αυτό. Αυτά από πλευρά μου. Αν έχετε ερωτήσεις, η διάθεσή σας ε, είμαι, αλλά ε, λέω να σταματήσω εδώ. Α, σήμερα επίσης αποφασίσαμε να μην κάνουμε τη συνεδρία συντονιστών γιατί δεν έχουμε τίποτα στην ημερήσια διάταξη. και ε, ίσως να κάνουμε άλλη μία συνεδρίαση μετά, ε, ε, πριν τα Χριστούγεννα. Θα δούμε τώρα γιατί είναι το θέμα του επιμερισμού των πόντων και θα, δούμε. Αυτά, Λαμπέρ. Είχε ζητήσει να μιλήσεις. Ευχαριστώ. Ναι. Θα δούμε ε, τι θα γίνει στη συνέχεια, όπως σωστά είπατε. Μιλήσατε ε, για την ε, τις επαφές που έχουμε με την ομάδα εργασίας για την πολιτική συνοχή. Όμως δεν θα έπρεπε να μιλάμε για την εφαρμογή, implementation. Νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Πρόκειται για τις ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Είπατε ότι ε, συμμετείχατε και στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υπάρχει μόνη πρόσκληση, υποτίθεται, από πλευράς της Προεδρίας, αλλά εγώ δεν έλαβα ποτέ πρόσκληση. Θα, ήθελα λοιπόν το Κοινοβούλιο να λαμβάνει με πάγιο τρόπο αυτές τις προσκλήσεις, όπως και στο παρελθόν. Κυρίως ε, και των αποφάσεων που λήφθηκαν την περασμένη εβδομάδα ε, διότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Είδα και το επίσημο ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσαν ικανοποιημένοι διότι έδωσε το Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του. Έτσι διάβασα. Νομίζω ότι κάτι μας διαφεύγει εδώ. Ή τουλάχιστον ε, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων δεν παρακολουθεί το ζήτημα όπως θα έπρεπε, διότι μιλάμε για το ζήτημα της περιφερειακής πολιτικής τα τελευταία 5-6 χρόνια. Νομίζω ότι ε, στις διοργανικές σχέσεις μας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη παρακολούθηση. Κάτι άλλο τώρα. Ο στόχος όλων αυτών που κάνουμε είναι εμπρόθεσμα να ε, ολοκληρώνουμε αυτά που μας έχουν ανατεθεί. Ε, παραδείγματος χάρη για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ξέρω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει εγκαίρως τις προσπάθειές μας, ε, αλλά με ποιο τρόπο αναρωτιέμαι, διότι ε, ε έχουμε καθυστερήσει ήδη και αν θέλουμε να ε, επιτύχουμε το στόχο μας ε, και δεδομένου το ότι πρόκειται για νομοτεχνική εργασία θα πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα. Ε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ξέρουμε για το θέμα των κλιματικών αλλαγών τι θα γίνει στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία ε, προκρίνει μια πράσινη προσέγγιση ε, Βεβαίω και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματευτούμε αυτό το ζήτημα. Ιδανικά θα ήθελα με τις συνεργασίες να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες μας. Αυτά τα σχόλια θέλω να κάνω προς το παρόν και από ό,τι φαίνεται είναι η επαύριο του... της επόμενης έκθεσης, της ε, μεγάλης μας εκδήλωσης, οπότε γυρνάμε στα συνηθισμένα. Πρόεδρος. Να απαντήσω στα σχόλια του συντονιστή του ΕΛΚΑ. Σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης θα κάνουμε τη συζήτηση στο 11, στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Θέλω καταρχάς να ακούσω τον εισηγητή, να δω πώς θα αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή. Επίσης να σας ενημερώσω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στην Ολομέλεια του Απρίλου. Αλλά καλύτερα να στοχεύσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Με την επιφύλαξη του Απριλίου, έτσι. Γιατί ανησυχώ. Γιατί ίσως να θυμάστε ότι το Συμβούλιο αρνείται τουλάχιστον για πέντε χρόνια, αν όχι περισσότερο, να δεχτεί τις α, τροπολογίες και να δεχτεί τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού. Τελικά φτάσαμε σε μια φάση όπου ε, έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Πολλά λοιπόν θα εξαρτηθούν από το πόσο θα απέχουμε από τη θέση του Συμβουλίου, πόσο θα απέχει το Συμβούλιο από εμά. Από αυτό εξαρτάται το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Εμείς θα πρέπει να στοχεύσουμε πάντως να οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία μέσα σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Θα γίνει η τελική παρουσίαση στις 18 Δεκεμβρίου και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Τον ε, Ιανουάριο θα έρθει και ο Έλληνας υπουργό και τότε μπορούμε στην Επιτροπή μας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι μόνο να συζητάω εγώ ας πούμε ως εκπρόσωπό σας ε, σε επαφή με τον εισηγητή. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ξέρω πάντως εδώ για τις προσκλήσεις προς το Συμβούλιο. Φυσικά η Προεδρία προσκαλεί. Συχνά όμως και συνάδελφοι που θέλουν να πάνε ζητούν να προσκληθούν. Και απλώς συνήθως η Προεδρία αντιδράει θετικά. Ρυθμίζουμε και τα ταξιδιωτικά έξοδα κτλ. Η Γραμματεία όμως δεν έλαβε κανένα αίτημα από κανένα. Πάντως η Προεδρία προσκάλεσε μόνο τον Πρόεδρο. Τώρα, για τους επόμενους μήνες, ε, ίσως θα έχει νόημα για την εφαρμογή να έχουμε μια ομάδα εργασίας ε, στο επόμενο, στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Άλλες ε, προτάσεις, άλλα σχόλια για τις ανακοινώσεις του Προέδρου, όχι. Πάμε στο σημείο 4 λοιπόν της μερικής διάταξης. Είναι η έκθεση της Ελίζα Σράντε. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για τις τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις της εγκατάστασης ευφυών δικτύων. Ελίζα, θα έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν, που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου για την έκθεση αυτή και που θα θελήσουν και στο μέλλον είναι συναρπαστική έκθεση. Είναι μια έκθεση για το μέλλον, για να επιλέξουμε νέες δυνατότητε στην περιφερειακή οικονομία και τον ιδεότερο ρόλο των ε, περιφερειών και των τοπικών φορέων ε, στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουμε ένα έγγραφο που ανέφερε και παραδείγματα. Είναι σημαντικό να σας θυμίσω ότι έχουμε μια σειρά παραδείγματα από την Αυστρία, από κάποια νησιά, ε, την Μαδέιρα, από το Χιχόν ε, στην Ισπανία, από την Ελλάδα <clears throat> και από την περιοχή Χάρτς στη Γερμανία, όπου περιφέρειες με ιδιαίτερα ευφυή τρόπο επιχείρησαν να προωθήσουν ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι αποκεντρωμένες είναι πηγές ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και προσπάθησαν να εξοικονομήσουν ενέργεια, να αναπτύξουν δηλαδή ένα σύστημα που θα τους επιτρέπει να επιτύχουν την ε, ενεργειακή αυτάρκεια. Υπενθυμίζουμε επίσης μία μελέτη που έγινε από την Κομισιόν πριν από μερικά χρόνια. Ήταν η μελέτη Περιφέρειες 2020. Ήταν ένα από τα πέντε κεντρικά σημεία. Έλεγε συγκεκριμένα ότι θα είναι η ενεργειακή εξάρτηση και ανεξαρτησία ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες. Δηλαδή, θέλουμε να διοργανωθεί αυτή η προσπάθεια έτσι, ούτως ώστε τα περισσότερα κέρδη να τα λαμβάνουν οι περιφέρειες και οι οργανισμοί τοπικής ε, αυτοδιοίκησης. Και διαπιστώσαμε ότι είναι βασικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης για την ανάπτυξή τους. Γι' αυτό αναφέρω για άλλη μια φορά τα παραδείγματα που αναφέρονται και εξηγούνται σε αυτό το έγγραφο εργασίας που, ήταν, ε, που είχε ως βάση μία έκθεση που είχαμε παραγγείλει εμείς ως Περιφερειακή Επιτροπή όπου αναφέραμε παραδείγματα βελτίστων πρακτικών. Αυτή η μελέτη για μένα είναι η βάση και της έκθεσης. Η έκθεση αυτή καθεαυτή αναφέρει πορίσματα. Δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει μετά τη μελέτη, μετά τα παραδείγματα, τι θα πρέπει να ακολουθήσει, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά στο μέλλον. Πρώτο σημείο, υπάρχουν νέες δυνατότητες για τις περιφερειακές οικονομίες, τις οικονομίες των περιφερειών. Υπάρχει ξαφνικά μια αλλαγή. Περιοχέ που ήταν απόλυτα εξαρτημένε, για παράδειγμα νησιά, που ήταν απόλυτα εξαρτημένε από το υπηρετικό μέρο τη χώρα όσον αφορά την ενέργειά του, μπορούν να αξιοποιήσουν ανασιώσιμε αποκεντρωμένε ενέργειε, ούτως ώστε όχι μόνο να έχουν ε, ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά μπορούν να γίνουν και παραγωγή και εξαγωγής ε, ενέργεια, δηλαδή να πουλάνε σε άλλε ε, περιφέρειες. Αυτό είναι μεγάλο κέρδο για τι περιφέρειες και ιδιαίτερα με περιοχές που δεν είχαν καμία δυνατότητα εισοδημάτων έχουν εδώ τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικοί οικονομικοί παίκτες στον τομέα αυτό. Για μένα αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα. Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι αυτή η δυνατότητα θα μπορέσει να αξιοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν οι συνθήκες πλαίσιο. Και αυτά είναι ιδιαίτερα τεχνικά θέματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συστήματα ούτως ώστε η ενέργεια να, να είναι αμφίδρομη. Δηλαδή ε, θα πρέπει, εάν θέλουμε να μπορούν να πουλήσουν ενέργεια οι ε, περιφέρειες, να υπάρχει το δίκτυο για να μπορούν να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Και οι περιφέρειες δεν θα έπρεπε να μπορούν να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια μόνο στο κεντρικό ε, δίκτυο, αλλά να μπορούν απευθεία να, ε, να παρέχουν αυτή την ενέργεια στους πολίτες της, της περιφέρειάς τους. Και αυτό θα οδηγήσει και σε εξοικονομήσεις ενέργειας που θα το συνδυάσουμε με φυσικά την ε, ανεξαρτησία. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει εμφυός. Για να γίνει εμφυός θέλουμε να υπάρχει η σωστή ε, τεχνολογία πληροφορικής και ε, τηλεπικοινωνιών. Διότι πέρα από το ενεργειακό δίκτυο, το δίκτυο πληροφορικής είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν αυτά τα ευφυή δίκτυα. Επιπλέον, αν θέλουμε να κερδίσουμε ενέργεια, ξέρουμε ότι για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Υπάρχουν περίοδοι όπου μπορεί κανείς να παράγει πολλή ενέργεια και κατόπιν πολύ λιγότερη. Υπάρχουν λοιπόν ε, μέγιστα και ελάχιστα παραγωγής. Και όταν έχουμε μέγιστο παραγωγής ε, μπορεί να μην χρειαζόμαστε τόση ενέργεια γιατί είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν ε, που παράγουν πολλή ενέργεια δεν τη χρειαζόμαστε και το χειμώνα αντίστροφα. Κεντρικό σημείο λοιπόν αυτών των ευφυών δικτύων είναι οι δυνατότητε αποθήκευση. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμη. Η έρευνα δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ούτως ώστε να έχουμε ιδιαιτέρως ευφυή αποθήκευση ενέργεια. Για παράδειγμα στη μελέτη αλλά και πέρα από τη μελέτη, έψαξα και γενικότερα, και έχουμε διαπιστώσει ευρύτερα στην Ευρώπη ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές. Δηλαδή αποθηκεύουμε ενέργεια ούτω ώστε μετά να την αξιοποιήσουμε στην λεγόμενη αϊ-κινητικότητα. Δηλαδή, πώς είναι η κατάσταση. Έχουμε την αναγκαία τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας, έχουμε την πληροφορική με τις, χωρίς την οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει το FES δίκτυο και μετά έχουμε και τις συγκοινωνίες. Διότι μπορούμε αυτή την ενέργεια που παράγεται να την αξιοποιήσουμε μέσω φόρτισης ε, μπαταριών για τα μέσα μεταφοράς και επίσης μπορούμε να την μεταφέρουμε και στα κτίρια μέσω ευφυών, ε, ε, δυνατοτήτων θέρμανσης για παράδειγμα στα κτίρια, γραφείων, σε σπίτια. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη εμπλέκονται τέσσερι τομεί. Αυτή η ιδέα λοιπόν των ευφυών δικτύων δεν είναι μόνο θέμα ενό δικτύου, δηλαδή φτιάχνουν ένα δικτύο και έγινε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. βεβαίω είναι στοιχείο κλειδί, είναι ολόκληρα συστήματα και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αν έχουμε αυτό το περίπλοκο σύστημα. Αυτό είναι κεντρικό σημείο τη έκθεση. Η οικονομική χρήση, το οικονομικό όφελο για τι περιφέρειε δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη συζήτηση για τα δίκτυα, θα υπάρξει αυτό το όφελος εάν καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ένα περίπλοκο σύστημα, να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα. Και στα προγράμματα που έχουμε γίνεται αυτή η προσπάθεια και κατόπιν έρχεται το οικονομικό κέρδος. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό πόρισμα. Το δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται απασχόληση. Γιατί θέσεις εργασίες που προηγουμένως ήταν αλλού, γιατί μόνο δέχονταν, ε, δέχονταν ενέργεια οι περιφέρειες, τώρα παράγουν ενέργεια, άρα υπάρχουν δουλειές. Στον τομέα εξοικονόμηση ενέργειας, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε ε, πολλά, ε, πολλές υποδομές, δεν είναι μόνο νέες θέσει εργασία που χρειάζονται νέες ειδικεύσεις, αλλά είναι και, για παράδειγμα, κατασκευές. Δηλαδή μόλις αρχίσει κάποια περιφέρεια να προσπαθεί να οικοδομήσει όλο αυτό το δίκτυο, δημιουργούνται θέσει εργασία. Το άλλο είναι πόσο σημαντικό είναι αυτά για τους πολίτες Αυτά τα συστήματα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εάν συμμετάσχουν όλοι σε μια περιφερεια. Αν υπάρχει ετοιμότητα από πλευρά των πολιτών να εισαγάγουν αυτό το σύστημα. Και ξέρουμε ότι οι πολίτες θα ε, δεχθούν να εισαγάγουν αυτό το σύστημα εάν δουν ότι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Γι' αυτό η συμμετοχή των πολιτών συγκεκριμένα και στα πρακτικά ωφέλη είναι κεντρικό στοιχείο για να δημιουργήσουμε την διάθεση των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτά τα ευφυή συστήματα. Ο ρόλος των πολιτών, η συμμετοχή, ο κοινός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός του πώς θα συμμετάσχουν, πώς θα κερδίσουν εάν θέλουμε ακριβώς να κερδίσουμε για παράδειγμα μέσω συστημάτων ε, ανεμογεννητριών είναι κεντρικό. Γιατί είναι κεντρικό και περνάω στο επόμενο γιατί είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για αυτά τα εφηδίκτια, είναι η προστασία των δεδομένων. Αν θέλουμε ένα ευφυές δίκτυο ούτω ώστε να έχουμε στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό χρειάζεται να συλλέξουμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική σφαίρα και πολύ βαθιά με την ιδιωτική σφαίρα. Άρα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Και γι' αυτό η προστασία των δεδομένων είναι κεντρικό σημείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χρειαζόμαστε συστήματα όπου με ανώνυμο τρόπο θα συλλέγονται αυτά τα στοιχεία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την έρευνα για αυτά τα FEE δίκτυα. Είναι η ανωνυμοποίηση των στοιχείων γιατί αλλιώ δεν θα συμμετάσχουν οι πολίτες. Επόμενο, το πλαίσιο για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Και το πλαίσιο πρέπει να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα επιδοτήσεις. Έχουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων που είναι αρκετά περιορισμένο διότι αντιμετωπίζει κάθε κλάδο και χωρισμένα. Αλλά είπα ότι αυτό το σύστημα θα λειτουργήσει μόνο εάν είναι διατομεακό. Εάν υπάρχει χρηματοδότηση για ε, πολλού τομεί μαζί. Αλλά αυτά δεν προβλέπονται. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα ευφυή δίκτυα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα επιδοτήσεων. Αυτό είναι ένα από... Αυτός είναι ένας από τους ε, δυσχερέστερους γόρδιους δεσμούς που πρέπει να λύσουμε αν θέλουμε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα επιδοτήσεων. Να φροντίσουμε δηλαδή να είναι δυνατόν οι περιφέρειες να μπορούν να φορτίζουν μπαταρίες και μετά να τις χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν τοπικές εγκαταστάσεις και υποδομή και διοίκηση που να μπορούν να διαχειρίζονται από κοινού όλους, όλους αυτούς τους τομείς. Όχι, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να κλείσουμε τις τοπικές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, οι τοπικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ε, λειτουργήσουν διατομέακα. Τελευταίο σημείο επ' αυτού. Χρειαζόμαστε διαμεθοριακή συνεργασία. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, μεθοριακές περιφέρειες οι οποίες είναι πολύ μακριά από τις κεντρικές περιοχές της χώρας τους, αλλά είναι πολύ κοντά σε άλλες περιφέρειες άλλων χωρών. Δηλαδή υπάρχουν ε, περιοχές ε, που και ιστορικά έχουν σχέσεις, αν και ανήκουν σε διαφορετικές χώρες, έχουν συνεργαστεί, θα μπορούσαν να αναπτύξουν κοινά συστήματα. Για τις επιδοτήσεις λοιπόν, έχουμε πει στην κατάσταση, θα ήταν καλό τέτοιες ε, διδημοποιημένες ε, μεθοριακές περιφέρειες να αναπτύξουν κοινά συστήματα. Αυτό μας θυμίζει την έκθεση για εκείνο τον κανονισμό του συναδέλφου Τσέλα που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει περιφερειακή συνεργασία για αυτά τα κοινά συστήματα. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε την αναγκαία όθηση, μόνο μέσω δημιουργίας οργάνων ευρωπαϊκής συνεργασίας όπως ε, αυτά που περιέχει το κανονισμός Τσέλα, περιέχονται στο κανονισμό Τσέλα. Αυτό είναι πολύ βασικό για τα FEE δίκτυα. Αυτό είναι βασικά το περιεχόμενο και τα απορίσματα της έκθεσης. Άλλα δύο όμως να αναφέρω. Το πρώτο, έγραψα την έκθεση αρχικά στα αγγλικά. Ήταν πολύ επιστημονικό και τεχνικό θέμα και είναι καλό οι τεχνικές έννοιες που ε, ε, περιέχονται. Ε, αυτές λοιπόν οι έννοιες είναι δύσκολο να τις μεταφράσω στα γερμανικά όταν προσπαθώ. Λοιπόν το πρωτότυπο είναι αγγλικά. Ε, κοίταξα τώρα τη γερμανική μετάφραση και υπάρχουν ε, αρκετά προβλήματα με την ε, μετάφραση ιδίως για αυτές τις τεχνικές έννοιες. Λοιπόν θα χρειαστεί να κάνω μερικές ε, τροπολογίες για να ε, λύσουμε αυτά τα προβλήματα γιατί αλλιώς ορισμένες έννοιες, ε, ορισμένες έννοιες βγαίνουν λάθος. Ε, θα κοιτάξουμε μετά και την, και την γαλλική μετάφραση να δούμε ότι τουλάχιστον αυτά οι τρεις μεταφράσεις είναι καλές. Δεν μπορώ να κάνω περισσότερα, τα πολωνικά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά το πρωτότυπο λοιπόν είναι αγγλικά, αν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα για τη μετάφραση, για αυτές τις τεχνικές έννοιες γιατί ορισμένε φορέ μεταφράζονται εντελώ διαφορετικά. Σα παρακαλώ, ε, ε, το πρωτότυπο είναι το αγγλικό. Νομίζω ότι ευχαριστούμε πολλέ τροπολογίε Και ο Πολωνός συνάδελφο έχει την εντύπωση ότι είναι ακατανόητα ορισμένα θέματα ε, στα πολωνικά. Και αυτό δεν είναι καλό γιατί είναι πολύ σημαντική για την Πολωνία αυτή η έκθεση. Σα παρακαλώ, κοιτάξτε λοιπόν με βάση τα αγγλικά τι θα μπορούσε να σημαίνει το πολωνικό κείμενο. Το δεύτερο, Η Επιτροπή Ήτρα με βάση τον κανόνα 50 συντάσσει μια έκθεση. Έχω συνεργαστεί στενά με τον ε, Σουηδό συνάδελφο που είναι εισηγητής. Έχουμε την ίδια γραμμή συνολικά και αυτή τη βδομάδα στην Ήτρε θα ψηφίσουν για την έκθεση αυτή. Και μετά η συμβολή τους θα έρθει να συμπεριληφθεί ως αυτόνομο τμήμα στην έκθεσή μας και θα πρέπει η Γραμματεία να κοιτάξει τι τροπολογίες της ήτρε θα πρέπει να ψηφίσουμε κι εμείς ή μπορούμε να τις αφήσουμε άλλες όπως είναι. Αυτό είναι τεχνικό θέμα. Λοιπόν, ε, άφησα στην Ήτρε τα τεχνικά θέματα και εγώ περιορίστηκα στα θέματα όπου πρόκειται για να δημιουργήσουμε οικονομικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας μέσω των ευφυών δικτύων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάν από το ΕΛΚΑ. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με τα τσέχικα, να μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα σας. Σας διαβεβαιώ ότι η μετάφραση προς τα τσέχικα είναι θαυμάσια. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, Είναι μια πολύ περιπλοκή κατάσταση εδώ. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτόν τον όρο. Τον συναντάμε τον όρο αυτό εφή δίκτυα παντού και ειδικά όταν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ασταθείς ε, ενεργειακές πηγές, ειδικά ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα διανομής ενέργειας. Και ομολογώ ότι Προσπάθησα να σκεφτώ λύσεις για το πρόβλημα. Μοιάζει άπιαστο αυτό το, το πρόβλημα, δηλαδή όλοι μιλάνε για αυτό, αλλά κανένας δεν το έχει δει απτά. Υπάρχουν στοιχεία των εφιών δικτύων που εφαρμόζονται σε διάφορα συστήματα διανομής, αλλά δεν υπάρχει πραγματικά ανεπτυγμένη έννοια ενός εφικτού, εφιούς δικτύου, ολοκληρωμένη με όλες τις διαστάσεις. Επίσης, το θέμα είναι περισσότερο ευνητικό ακόμα, παρά κάτι που είναι πραγματικότητα. Έχουμε βεβαίως μπαταρίες, οι οποίες καλές είναι. Έχουμε παραγωγή από νερό, χρησιμοποιώντας το υδρογόνο αλλά όλα αυτά τα μέσα δεν είναι κατάλληλα για τη βιομηχανική χρήση. Δεν αρκούν για τις βιομηχανίες αυτές οι μορφές ενέργειας. Αυτά ήθελα να πω για τα e δίκτυα. Τώρα, η προσέγγιση της εισηγήτριας. Ποια είναι. Αυτή επικεντρώθηκε σε ένα στοιχείο, το οποίο είναι ακριβώς αυτά τα περιφερειακά ευφυή e δίκτυα ή μάλλον ε, περιφερειακά εφή συστήματα παραδίκτυα. Όταν υπάρξουν αυτά τα συστήματα, όταν και όποτε. Θα ήθελα η Επιτροπή να αναλύσει πόσο θα κοστίσουν οι επενδύσεις ε, σε αυτά τα εφή συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Τα νούμερα που έχουμε λάβει που έχουν διαρρεύσει καλύτερα είναι εντυπωσιακά. Φυσικά υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία ακούγονται ξανά και ξανά, αλλά πρέπει να δούμε και το κόστος όλης αυτής της ιστορίας. Το πιο καλό πράγμα που εμπεριέχει η έκθεση, η οποία γενικά είναι θαυμάσια και σοβαρή, είναι το κομμάτι που αφορά την προστασία των δεδομένων. Αν είναι να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα, τότε πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τα νοικοκυριά, αν όχι τα άτομα και τις συνήθειές τους. Και αν τα δεδομένα αυτά πέσουν σε λάθος χέρια, αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Επομένως, είναι απόλυτα αναγκαίο να επιλύσουμε καταρχήν αυτό το θέμα. Και θεωρώ ότι μας προειδοποίησε επαρκώς, με πολύ σοβαρό τρόπο, η συγγήτρια γι' αυτό. Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα που κατά την απόψή μου είναι λίγο αμφιλεγόμενα. Αυτό που ζητάει δηλαδή για δεσμευτικούς στόχους μέχρι το 2030 για την, ανεώση, την αποτελεσματικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις εκπομπές. Αυτά είναι θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί, συζητιώνται ακόμα. Δεν ξέρω αν πρέπει τελικά να υποβάλω τροπολογίες για αυτά τα θέματα για να έτσι μαλακώσουμε λιγάκι αυτό το τμήμα του κειμένου. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές θετικές επιπτώσεις στη λεγόμενη αγορά εργασίας, νομίζω ότι η μεγαλύτερη επίπτωση των φωτοβολταϊκών, ας πούμε, ε, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, θα είναι στην Κίνα. Δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξο λοιπόν, τόσο υπεραισιόδοξο, παρότι σίγουρα κάποιες θετικές επιπτώσεις στην περιφερειακή αγορά εργασίας θα υπάρξουν. Δεν θα είναι εντελώ άνευ επιπτώσεων αυτή η ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας βάσης για την ανάπτυξη αυτών των θεών δικτύων, εκεί συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι χρειαζόμαστε αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, παρότι πρέπει να προχωρήσουμε με σοφροσύνη. Και θα ήθελα ακόμα μια φορά να σας υπενθυμίσω την ε, ιστορία των βιοκαυσίμων, όπου ήμασταν υπεραισιόδοξοι. Και στο ενεργειακό μείγμα υπάρχει μόνο 10% βιοκαυσίμων και όλοι ξέρουμε τι κατάληξη και αυτή η ιστορία. Επίσης, δεν θα ήταν καλό να επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε με την ηλιακή ενέργεια που νομίζω ότι μείωσε την ανταγωνιστικότητά μας. Επομένως, ε, έξυπνα δίκτυα, ναι. Περιφερειακή ανάπτυξη, ναι. Αλλά θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις πιθανές ε, επιπτώσεις. Από τους σοσιαλιστές. Καταλήνα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Σόντερ για την ε, ε, διαθεσιμότητά της για να συνεργαστούμε. Ήδη μέσω του εγγράφου εργασίας συνεργαστήκαμε και στόχος μας είναι φυσικά να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος γιατί θέλουμε επίσης να αυξήσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά θα τα επιτύχουμε μόνο εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από οποιοδήποτε τομέα είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν γιατί βλέπουν ότι ωφελούνται. Τέθηκε ένα αμφιβόλο εάν αυτό μπορεί να γίνει. Δεν ε, θα ήθελα να ε, το αμφισβητήσω αυτό γιατί έχουμε μια περιφέρεια, το Burgenland στην, ε, στην Αυστρία, που είναι η πρώτη περιφέρεια που ενώ πριν από 15 χρόνια δεν παρήχε καθόλου ρεύμα, τώρα το φθινόπωρο κατάφερε να καλύψει με δική της ενέργεια όλες τις ανάγκες και του χρόνου ή σε δύο χρόνια θα είμαστε και πολιτές ενέργειας. Αυτό γίνεται λοιπόν σε μια περιφέρεια της Ένωσης όπου για πρώτη φορά το 1997 όπου πήραμε κάποια χρηματοδότηση συνολικά λάβαμε 100 εκατομμύρια από τα διαθρωτικά ταμεία. Στην αρχή δημιουργήσαμε πάρκα ανεμογεννητριών, όπως είπε η κυρία Σρέντερ. Έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και σε παραδοσιακούς τομείς, κατασκευές για παράδειγμα. Έχουμε χιλιάδες απασχολούμενους, ε, είχαμε μάλλον όταν φτιάχναμε αυτά τα πάρκα και φτιάξαμε, ε, στήσαμε πάνω από 300 ανεμογεννήτριες. Οπότε έχουμε οικονομική αλλά και οικολογική αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήσαμε 1.260.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Με αυτή την ε, προσπάθεια επίσης έγινε και μια ανώτερη σχολή στην περιοχή μας που εκπαιδεύει νέους ανθρώπους για να εργαστούν σε αυτό το τομέα λέγεται ανώτερη σχολή για τεχνική ανανεώσιμων ανεμογεννήτρες. Αυτό είναι πολύ καινοτόμο. Στην περιοχή μας, στο Ομοσπονδιακό κράτος Μπουργενλάντ, έχουμε 160 ε, νέες θέσεις εργασίας που καλύπτονται από αποφύτους αυτής της σχολής. Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτά τα ευφύ συστήματα μπορούμε στο μέλλον να έχουμε και οικονομικά αλλά και οικολογικά βιώσιμα αποτελέσματα. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η έκθεση, διότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε όχι μόνο ε, τα δίκτυα αλλά και τις δυνατότητες αποχύτευσης, είναι πολύ σημαντικό. Και έχω κάποιες επιφυλάξεις, αναφέρθηκε ήδη, ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει όλα αυτά μόνο εάν καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν και επίσης εάν επιτύχουμε τη σωστότερη δυνατή λύση για την προστασία των δεδομένων. Γιατί αλλιώς αυτή η, αυτή η μετάβαση από την κεντρική παραγωγή στην αποκεντρωμένη ε, παραγωγή ενέργειας δεν θα περάσει τον πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φανίστε λόγω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω και εγώ αντίστοιχα σχόλια να κάνω. Συμφωνώ γενικά με την ε, έκθεση και τις ιδέες, δηλαδή να τονώσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να αναπτύξουμε μια οικονομία ουδέτερη σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, χάρη στα ευφύ δίκτυα και μια ευφύ ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές περιφερειακές πτυχές στην έκθεση. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία που θα ήθελα να πω. Μιλάμε για δεσμευτικούς στόχους στην έκθεση. Για αυτό το θέμα ξέρετε ότι κάναμε έντονες συζητήσεις. Επίσης υπάρχει μια σύσταση να περάσουν τις κρατικές ενισχύσεις σε άλλες μορφές ενισχύσεων. Ας το σκεφτούμε αυτό το θέμα. Μπορείς να δώσεις κίνητρα στην έρευνα πριν περάσει στο εμπόριο, αλλά για να εγκαταστήσουμε έξυπνα δίκτυα, αυτό είναι θέμα της ελεύθερη αγορά, Ας το αφήσουμε στην ελεύθερη αγορά, να παίξει το ρόλο της. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και το κοινό συμφέρον αυτών των προγραμμάτων. Αυτή η διατύπωση όπως υπάρχει τώρα στο κείμενο είναι πάρα πολύ γενικόλογη. Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, για την ε, για την ανάθεση των ε, συμβάσεων. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη φρασιολογία. Επίσης υπάρχουν και πολιτικά θέματα τα οποία θα πρέπει να απεικονίζονται στην έκθεση. Πέραν τούτου, γενικά συμφωνώ με την έκθεση, η οποία είναι πολύ εμπεριστατωμένη, πολύ ενδελεχής. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, ευφυή εξειδίκευση τη βάζουμε παντού αυτή τη λέξη, αλλά βλέπουμε ας πούμε ότι στη Γερμανία εκπαιδεύουμε νέους ε, μηχανικούς για αυτό τον τομέα. Στη χθεσινή συνάντηση ήρθε ένας εκπρόσωπος από την Ολλανδία και μίλησε για την ενεργειακή αξία και για την ε, διανομή φυσικού αερίου. Αλλά δεν θέλουν απλώ να εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο, θέλουν ε, να συνεργαστούν με άλλες περιφέρειες ε, ε, που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Επομένω, θα έχουμε και ανταγωνισμό, θα έχουμε συνεργασία μεταξύ των περιφερειών που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το, το θέμα και να δώσουν μια ευκαιρία στα έξυπνα δίκτυα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους νέους κανονισμούς για να δώσουμε κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη συνεργασία των περιφερειών. Ίσως η Ήτρε θα ασχοληθεί, δεν ξέρω, δεν είναι και πολύ σαφές ακόμα. Ποιοι τομεί είναι τη σίτρε και ποιοι τομεί είναι τη Ρέτζι, δεν ξέρουμε ακριβώ. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι για να ξέρουμε και σε τι θα ψηφίσουμε. Υπάρχει το πρόγραμμα Ορίζοντα και υπάρχει και ένα ειδικό τμήμα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας. Και υπάρχουν τέσσερα σημεία σχετικά και ένα από αυτά μιλάει ακριβώς για τα ευφύ δίκτυα. Ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί έχουμε ήδη πέντε κέντρα στην Ευρώπη που ασχολούνται με τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα. Έχουμε δηλαδή το ερευνητικό κέντρο, το κέντρο κατάρτισης, θα πρέπει δηλαδή όλες αυτές τις αρμοδιότητες να τις διασυνδέσουμε με τα τέσσερα σημεία που αναφέρει το κείμενο για την ενέργεια. Η έκθεση αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, λοιπόν, για να επηρεάσουμε τα πράγματα, να έρθουμε σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να διασυνδέσουμε διαφορετικούς στόχους, να τους βάλουμε σε ένα πλαίσιο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά όπως είπε και ο Γιάνν, θα υπάρξουν και προβλήματα. Είτε μιλάμε για την, τις είτε μιλάμε για την ηλιακή ενέργεια, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να τα διασυνδέσουμε, να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο και ο καταναλωτής να γίνει πιο ανεξάρτητος. Να λέει, ας πούμε, δεν θέλω αυτή την μορφή ενέργειας, γιατί δεν την παράγει ας πούμε το κτίριό μου ή η περιοχή μου ή η περιφερειά μου. Θέλω την άλλη. Αυτό μπορούμε να ενθαρρύνουμε και εδώ μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας και να δούμε και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έχουμε έξι μήνες για τις εκλογές, μπορούμε να, τις αξιοποιήσουμε αυτούς τους μήνες. Έχουμε μια καλή ευκαιρία λοιπόν και σας ευχαριστώ για την έκθεση. Ευχαριστούμε ε, ευχαριστούμε πολύ την Ελίζα Πατρισφέντερ για την έκθεση και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Φυσικά είναι κατανοητό για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, για τα ε, οικονομικά στοιχεία, την απασχόληση. Ε, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας ως Επιτροπή, για αυτό που συζητάμε, το αντικείμενό μας, δηλαδή την περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική ότι η έκθεση γίνεται σε αυτή την Επιτροπή τώρα. Να πω δύο λόγια ότι ακόμα και αν είχαμε δυσκολία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έπρεπε να επιταχύνουμε τη μετάβαση, ακόμα και αν ήταν πιο ακριβές, κάτι που δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό πλέον, γιατί αυτά που βλέπουμε έχουν τεράστιο κόστος το οποίο δεν το έχουμε υπολογίσει. Η καταστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Φιλιππίνες, Σαρδινία και τελευταία και σε ένα νησί στη χώρα μου, στη Ρόδο, ε, είναι τεράστιο οικονομικό κόστος. Δεν το υπολογίζουμε όταν συζητάμε για το κόστος των ανώσιμων πηγών ενέργειας ή των επενδύσεων. Ε, άκουσα ότι το κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες από την καταστροφή τώρα ήταν 35 δις. Ε, 10 δις Φιλιππίνες κλπ. Αλλά υπάρχουν και τα χιλιάδες θύματα, δηλαδή ακόμα και αν δεν είχαμε καμία οικονομική καταστροφή. Άρα είναι πιο ευφυές να επενδύουμε στην καινοτομία, στην ανάπτυξη νέων λύσεων, αντί να πληρώνουμε το κόστος, όπως έχει πει και η έκθεση Στέρν της κλιματικής αλλαγής. Άρα το κόστος είναι πάντα σχετικό, είναι πώς θα το προσεγγίσουμε. Αλλά πιστεύω το πιο σημαντικό είναι ότι ε, αλλάζει πλήρως το ενεργειακό μοντέλο και η έννοια περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί μέσω των ευφυών δικτύων, το αναφέρει πολύ αναλυτικά η έκθεση, στην πραγματικότητα μπορούμε να παράγουμε και στον πιο μικρό τόπο την ενέργεια που χρειάζεται, που σε πολλές περιπτώσεις σήμερα είναι εισαγόμενη. Σα αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για τα δημοσιονομικά. Στα νησιά που είμαι εγώ στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, το κόστος μόνο του πετρελαίου το οποίο εισάγεται κάθε χρόνο για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες είναι 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αν κάθε χρόνο επενδύαμε 700 εκατομμύρια, θα είχαμε πολύ περισσότερους πόρους από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη αυτών των ευφυών δικτύων, γιατί μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαφορετικά ε, μοντέλα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως να τα συνδέσουν με παραγωγικούς τομείς όπως είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές, ακόμα και η ναυτιλία, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη οικονομική σημασία αλλά και δημοσιονομική σημασία. Η, η, η Τρόικα θα έπρεπε αυτά που στάμε εδώ να τα βάζει στην ατζέντα της και να βοηθάει τις χώρες να τα αξιοποιήσουν. Δηλαδή αντί να λέει κόψτε 700 εκατομμύρια από τις συντάξεις και από τους μισθούς, θα έλεγε επενδύσει 700 εκατομμύρια για εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνα δίκτυα. Είναι ο διαφορετικός τρόπος, νομίζω, εφαρμογής. Ε, και κυρίως αυτό που δίνει τη δυνατότητα, μια τέτοια στρατηγική, είναι να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών. Δηλαδή υπάρχουν περιφέρειες που είναι μειονεκτικές, γιατί αναγκάζονται να πληρώνουν τα πάντα για να τα εισάγουν. Τρόφιμα, ενέργεια, ε, συνδέσεις ναυτιλιακές με τα ευφυή δίκτυα μπορούν να γίνουν παραγωγή και εξαγωγή. Δηλαδή να φορτίζουν ένα πλοίο το οποίο θα βασίζεται εν μέρη και στη χρήση ανώσιμων πηγών ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να βοηθήσουμε να το συνδέσουμε με τα ναυπηγεία που είναι σε κρίση, με τα μεταφορικά συστήματα κτλ. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Ε, ένα πολύ σημαντικό όμως είναι να βοηθήσουμε εν ώψη και του 2014-2020 τις περιφέρειες να ενημερωθούν και να κάνουν το σχεδιασμό. Πολύ σωστά λέει η Ελίζαμπεθ ότι πρέπει να κάνουν σχέδια, αλλά πρώτα πρέπει και να το ξέρουν το αντικείμενο. Πολλές περιφέρειες είναι προχωρημένες, όπως αναφέρθηκαν παραδείγματα, αλλά άλλες περιφέρειες έχουν πλήρη άγνοια ακόμα και για τον όρο εφηδίκτια στα θέματα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε γρήγορα ένα τρόπο ε, τέτοιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Και ένα τελευταίο, Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις και το αναφέρει σαφώς η έκθεση της Ελίζα Μπεθ, λέει ορισμένε κατηγορίε δημοσίων και κρατικών ενισχύσεων να θεωρούνται συμβατέ με την εσωτερική αγορά. Δεν πάει η αγορά παντού για να αναπτύξει τα δίκτυα. Σκεφτείτε ότι πάρα πολλέ ορεινέ και νησιωτικέ μειονεκτικέ περιοχέ δεν πρόκειται ποτέ να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το χάσμα του με άλλε περιφέρειε, αν περιμένουν από την αγορά να το κάνει αυτό. Επομένω, να μια κατηγορία νησιωτικών, νησιωτικέ και ορεινέ απομακρυσμένε μειονεκτικέ περιοχέ που εκεί πράγματι μπορεί να ισχύσει αυτή η συνθήκη. Α τι περιγράψουμε. Α τι περιγράψουμε, αλλά προφανώ σε μια αναπτυγμένη περιφέρεια δεν χρειάζεται ίσω γιατί θα βρεθούν και ιδιωτικοί πόροι και δημόσιοι πόροι. Αλλά α προσδιορίσουμε και να πούμε ιδιαίτερα για νησιωτικέ ορεινέ μειονεκτικέ περιοχέ, θα πρέπει να θεωρείται αυτό ότι είναι συμβατό με του όρου ε, της εσωτερικής αγοράς. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρίγκα, από την... η κυρία Σκαρίγκα διορθώνει πρόεδρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση για την ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και έχουμε και ένα συνάδελφο από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ενέργειας ε, που μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα. Ε, από πλευράς Επιτροπής συμφωνούμε ότι είναι κέριος ρόλος των περιφερειών και των πόλεων για να επιτύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους και όντως όπως αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης θα χρειαστεί μετεξέλιξη του ενεργειακού συστήματος που θα αντιληφθεί ακριβώς ως ένα συνολικό σύστημα. Χρειάζεται οι καινοτομίες, ε, όπως σωστά μα είπε και η συγγήτρια. Λοιπόν, στα πλαίσια της στρατηγικής ε, θα ε, εντατικοποιηθούν οι επενδύσεις και ως προς την αποτελεσματικότητα των ανανεώσιμων και ως προς τα ευφυή e e δίκτυα, το συνολικό σύστημα καθώς και την έρευνα και την καινοτομία για αυτό το ζήτημα. Ε, για τα εφή e e δίκτυα, όπως αναφέρθηκε, ε, αναμένονται σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις ε, φυσικά Οπότε θα συστήναμε να χρησιμοποιήσουμε χρηματοπιστωτικά εργαλεία, να συνδυάσουμε εγγυήσει, ε, δάνεια, ε, ε, κινητές αξίες, ομόλογα. Με έναν πολύμορφο σχεδιασμό θα μπορούσαμε να επιτύχουμε σημαντικές ιδιωτικέ επενδύσεις με την υποστήριξη φυσικά και του δημοσίου τομέα. Όπως ακούσαμε, φυσικά είμαστε σε ένα πρόωρο στάδιο όπως τόνισε και ο κύριος Φανίστερο για τα FEE δίκτυα και θα έπρεπε να αναπτύξουμε περαιτέρω κάποια πιλωτικά προγράμματα που θα λειτουργήσουν ως υποδείγματα για να έχουμε κάποια πρότυπα στον τομέα αυτό ώστε να αρθούν ε, τεχνικές και μη ε, δυσκολίες ε, που παρεμποδίζουν περαιτέρω ανάπτυξη προς το παρόν. Κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και χρήσιμη αυτή η έκθεση για τις ε, περιφέρειες, ε, κυρίως όταν δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, διότι βλέπουμε ποιες εμπειρίες ήδη υπάρχουν και αυτό αποτελεί πηγή έμπνευση ε, για τις ε, περιφέρειες ε, για να συνειδητοποιήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια χρηματοδότηση. Επίσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελα να προσθέσω ότι έχει γίνει μια μελέτη και στο κοινό ερευνητικό κέντρο υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης όπου μπορείτε να δείτε τι έχει γίνει στον τομέα αυτό στα διάφορα μέρη της Ευρώπης. Κατόπιν, ε, ο εξυγχρονισμό των κρατικών επιδοτήσεων είναι ένα άλλο ε, στενά συνδεδεμένο ζήτημα. Όπω σωστά αναφέρει η έκθεση, οι μελλοντικέ κατευθυντήριε γραμμέ ε, για τι κρατικέ ενισχύσει στον τομέα του περιβάλλοντο ακόμη τώρα ε, τι επεξεργαζόμαστε. Συνεχίζει τη διαβούλευση και φυσικά θα λάβουμε υπόψη την συμβολή σας πρωτού ολοκληρώσουμε τη μελέτη και καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Ξέρετε ότι αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, συνεχίζονται και όπως ε, σωστά είπε ο κύριος Χρυσόγελος, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στις περιφέρειες, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής με τρόπο ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Σας ευχαριστούμε για την έκθεση και δίνω το λόγο τώρα στον συνάδελφο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαρι... Γιάννη Πάνικ λέγομαι και είμαι προιστ ενό ε, του τμήματο ε, που ασχολείται με τα ΕΦΗ, δείκτε στη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία. Φυσικά, όπω σωστά τονίσατε κι εσεί, υπάρχουν διάφορα προγράμματα ΕΦΗΟΝ δικτύων που ε, λειτουργούν και ήδη επενδύονται κονδύλια σε αυτέ τι ΕΦΗ τεχνολογίε. Δεν νομίζω ότι θα ήταν ακριβέ να πούμε ότι είναι μία όαση προ το παρόν τα ΕΦΗ δίκτυα, που κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί. Όχι, μπορούμε ήδη να καταδείξουμε ότι λειτουργούν λειτουργούν στην πράξη σε περιφερειακή βάση. Συμφωνώ βεβαίω ότι αυτό δεν επαρκεί και πόρο απέχουμε και δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω ε, η ιδέα, αλλά αυτό δεν μα εμποδίζει από το να αναγνωρίζουμε την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και από αυτού να χτίσουμε τι προσπάθειε μα ε, διότι χρειαζόμαστε τα υφή στην Ευρώπη. Νομίζω στη σημερινή συζήτηση μεταξύ άλλων βλέπουμε συγκεκριμένα ωφέλη, βλέπουμε ε, και στην καθημερινή καθημερινή ζωή. Το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, είδαμε τη ζημιά ε, που μπορεί να προκληθεί εάν τα υφή δίκτυα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ουσιαστικά τη καθημερινή ζωή, ε, μεγάλε ε, φυσικέ καταστροφέ ή άλλε πηγέ ανισορροπιών που προέρχονται από την αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υποστηρίζω λοιπόν τις δηλώσεις των μελών της Επιτροπής σας. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ δύο παρατηρήσεις ε, που θα θέλαμε να τονιστούν ότι περαιτέρω μέσα στην έκθεση. Πολύ καλό που τονίζεται η σημασία και η πρόκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσα στην έκθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, δεν πρέπει να παραγνωριστεί η σημασία του και είναι στοιχείο κλειδί για την εξέλιξη των εφιών δικτύων, αλλά ταυτόχρονα οι πολίτες θα πρέπει να δουν τα ωφέλη, η διεισόμαση, όχι μόνο να συμμετάσχουν και να θεωρηθούν ότι εμπλέκονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όμως να δουν δουν και απτά ωφέλη ε, των συστημάτων που τους προτείνονται. Από αυτή την ε, σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να ε, καθησυχαστούν ότι προστατεύονται τα δεδομένα, αλλά να γνωρίζουν, να έχουν πλήρη ενημέρωση σε σχέση με τη μελλοντική χρήση των δεδομένων και να γνωρίζουν τι είδους δεδομένα, ποια ακριβώς δεδομένα θα πάνε σε, ε, ε, ε κάποιες αρχές και να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι αρχές, ε, διότι πέρα από το διαχειριστή του δικτύου, ε, τα δεδομένα του κάθε καταναλωτή, του κάθε πολιτή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δίνει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για κάποιους άλλους ε, ε, φορείς ε, πέραν από το διαχειριστή του δικτύου δηλαδή όπως ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς επίσης τα συστήματα μέτρηση είναι πάρα πολύ σημαντικά η έκθεση μιλάει και τονίζει για την συστημική προσέγγιση όμως δεν αναφέρονται καθόλου δεν αναφέρεται το ακρογωνιαίος λήθος του εφιούς δικτύου που είναι το σύστημα μέτρησης, εφιές σύστημα θα πρέπει ε, οι ευφυείς μετρητές ε, να αναγνωριστούν ω τέτοιοι μέσα στην έκθεση. Δηλαδή βλέπουμε μέσα στην έκθεση των κρατών μελών ε, ότι η ανάπτυξη των ευφυών μετρητών είναι μια πραγματικότητα, όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές και όχι μόνο στα κράτη-μέλη. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, κάνουμε συγκριτικές μελέτες ε, που θα τονίσει τη σημασία ε, τη εφιούς μέτρηση. Χρειαζόμαστε όμω τη δική σα υποστήριξη και φυσικά την υποστήριξη του Συμβουλίου. Τελευταία παρατήρηση είναι ξεκάθαρο μέσα στην έκθεση ότι όχι μόνο τα κράτη, δεν πρέπει να εμπλέκονται όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και ε, οι περιφερειακέ κυβερνήσει, γιατί είναι και τα διαρθωτικά ταμεία. Πρέπει να κατέβουμε όμω και στο επίπεδο των τοπικών κυβερνήσεων, τη τοπική αυτοδιοίκηση, διότι και ο δικό του ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε έτσι ένα σημαντικό εργαλείο ε, διότι έχουμε το Covenant of Mayors, ε, το Σύμφωνο των Δημάρχων, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για τη συνεργασία και διοργανική συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το μήνυμα των ευφυών δικτύων να περάσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, οι τοπικέ κοινότητε και όχι μόνο οι περιφέρειε θα δουν τα ωφέλη των ευφυών δικτύων και θα θεωρήσουν ότι εμπλέκονται στην περαιτέρω πρόθεσή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ελίζαμπεθ, δύο λεπτά δεν μπορώ παραπάνω, διότι ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο μα και τρώμε χρόνο την επόμενη έκθεση. Σε παρακαλώ συνοπτική. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτον, για τις θέσεις εργασίας. Η εγκατάσταση ηλιακών εγκαταστάσεων δεν το εξήγησα σαφώς δεν είναι ότι θα, δημιουργήσει τόσο πολλές θέσεις εργασίας, ε, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται θέσεις εργασίας για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και κυρίως τον τομέα της πληροφορικής που ελέγχει όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, είναι ο τομέας κατασκευής, ο τομέας πληροφορικής, ο τομέας της μηχανολογίας για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ε, έχουμε μετά τη συντήρηση, τις επισκευές, επίσης την εγκατάσταση των ε, σωμάτων θέρμανσης και τα λοιπά, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι κλασικές περιφερειακές θέσεις εργασίας που ήδη περιφερειακά ε, καλύπτονται αλλά χρειάζεται κατάρτιση και ευχαριστώ την κυρία Κάτνμπαχ για την πρόταση να πω περισσότερα για αυτό το θέμα. Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι η μόνη πηγή ενέργειας. Υπάρχει η θέρμανση από τη γη, η θερμότητα από τη γη. Επίσης έχουμε και υδροελεκτρική ενέργεια, έχουμε και μικρές υδροελεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και από περιφέρεια σε περιφέρεια είναι εντελώ διαφορετικές πηγές ενέργειας. Όλες αυτές οι ανανεώσιμες βοηθάνε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που κατέθεσε σαφές ότι πρέπει να ακολουθήσουμε νέες μεθόδους και ότι είναι θαυμάσια τα παραδείγματα. Τόσο θαυμάσια που αξίζει να γίνουν ευρύτερα γνωστά, ούτως ώστε να συμμετάσχουν όλοι. Είναι σωστό ότι κυρίως επενδύει ο ιδιωτικός τομέας αλλά ευχαριστώ την Κομισιόν που κατέστησε σαφώς, σαφές ότι και ο δημόσιος τομέας έχει δυνατότητες να δώσει επιδοτήσεις που θα πρέπει να είναι μια όθηση. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η μεγάλη έκκληση για τον τομέα των επιδοτήσεων, τους ώστε να είναι αποδεκτές οι συνδυασμένες επιδοτήσεις, οι, διατομια... οι διατομιακές επιδοτήσεις, για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας. Ευχαριστώ τον Λάμπερτ για την ε, έννοια της εφιούς εξειδίκευσης που ανέφερε. Βεβαίως, ε, συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ την Κομισιόν που έθεσε το θέμα των ελέγχων από τους πολίτες. Να κοιτάξω τι άλλο έχω γράψει. Βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το τμήμα και βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είμαστε σαφέστεροι. Βεβαίως και οι ευφυείς μετρητές. Βεβαίως. Πολύ βασικό θέμα. Αλλά σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα της Ήτρε. Γι' αυτό το βγάλαμε εμείς. Είναι απάντηση και στην ερώτηση τι κάνει η Ήτρε. Αλλά θα κοιτάξω σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει, εάν έχουν θέσει τα θέματα αυτά εντός, γιατί και αυτοί θέλουν τους συμβασμούς τους. Εάν μέσω των συμβασμών των δεν καλύπτεται σαφώς, τότε θα το επαναφέρουμε εμείς το θέμα. Και οπωσδήποτε θα επιμείνουμε και στην Ολομέλεια μέσω τροπολογιών. όλα αυτά τα τεχνικά θέματα δεν τα ανέφερα εκπεφρασμένα, αλλά αυτό το έκανε επίτηδες. Αλλά τονίζω ότι αν η Ήτρε δεν τα συμπεριλάβει, τότε θα φροντίσουμε εμείς. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Νομίζω ότι θα είναι λόγω της κοινή εργασίας, θα είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα και ελπίζω ότι και είμαι πεπισμένο ότι θα συνεχίσουμε επιτυχώς εργασία μας. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό λοιπόν που έχεις αυτή την αντιμετώπιση ως εισηγήτρια. Ε, και να σας ενημερώσω ότι έχουμε στείλει την έκθεση εκ των προτέρων στους Κιώδης και στους Συμβούλους, ε, διότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για τις τροπολογίες. Αύριο στις 12 εκπνέει η προθεσμία, διότι προθέμεθα να, το, να ψηφίσουμε την έκθεση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Αυτά πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε και τα αποφασίσαμε. Περνούμε τώρα στο σημείο 5 ε, της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Σας ε, προετοιμάζω ψυχολογικά. Η Ελισμπιέτα Καταρζίνα Λουκασκέστια θα μας μιλήσει για την κοινή επιχείρηση σχετικά με τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους ε, ε, όλος ιδιαίτερος τον κύριο Λάμπερς, τον συντονιστή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας εκπροσωπεί στην Επιτροπή Βιομηχανίας, διότι Πιστεύω και ελπίζω ότι όλες οι συστάσεις μας ε, θα εγκριθούν από την ε, ε, Ήτρε. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην οποία, στις να αντεπεξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενέργεια και κυρίως η απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Ε, βεβαίως με τα νέα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να αναλυφθούν και νέες πρωτοβουλίες ε, για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Χρειαζόμαστε μία ε, βιομηχανία που βασίζεται στα βιοπροϊόντα. προϊόντα. Ε, ποιος είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης. Λοιπόν, ε, ε, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί σύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων με τρόπο ώστε να ε, δημιουργηθεί μια κοινή επιχείρηση η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από όλους όσους την ιδρύσουν. Για τους πόρους από το 2014 έως το 2020 διαθέτουμε ένα δις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι τρία δις από μια σύμπραξη. Ε, κοινοπραξία, συγγνώμη, όχι σύμπραξη. Ε, ποια θα είναι αυτή η κοινοπραξία, θα είναι μία μη εμπορική κοινοπραξία που ε, θα αξιολογήσει την αξιακή αλυσίδα για την ε, βιομηχανία των βιοπροϊόντων, μικρά κλάστερς, επιχειρήσεις, πλατφόρμα για την πληροφορική, ο, διάφορες οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να προσχωρήσουν σε αυτήν την κοινοπραξία. Προς το παρόν έχουμε 60 ε, ενδιαφερομένους, ε, KLM, Unilever, ε, έχουμε ερευνητικά Ινστιτούτα, πανεπιστήμια, startup επιχειρήσεις που ασχολούνται με ενεργειακά προϊόντα, είναι προφανές ότι αυτού του είδους η συνεργασία θα μας βοηθήσει ώστε να υπερπηδήσουμε τα οικονομικά προβλήματα. Όμως ε, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό διότι ε, αυτό το εγχείρημα είναι μια καταπληκτική πηγή καινοτομία. Η αξία ε, θα υπερβεί τα 200 δις μέχρι το 2020 ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχολήσεως και δημιουργία νέων προοπτικών για τις περιφέρειες και τις, κυρίως για την Ήπεθρο. Ε, ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι, όπως σας είπα, η ίδρυση μιας κοινή επιχείρησης που βασίζεται σε μια νέα σχέση ε, συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα ε, που εν μέρει χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της παραγωγής καινοτόμου ενέργειας αλλά και για την ε, κατασκευή νέων καταναλωτικών ε, προϊόντων ε, που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από την ευρωπαϊκή βιομάζα. Δημιουργία επίσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα ενισχύσουν τον επιχειρηματικό κόσμο σε όλα τα επίπεδα, από τις προμηθευτές βιομάζας, γεωργούς, εγκαταστάσεις βιοδήληση, καταναλωτές. Στη συνέχεια θα τονωθούν διατομιακές σχέσεις, όπως σας έλεγα και στην αρχή, ε, θα εγκατασταθούν ε, νέες ε, συγγνώμη, θα δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις σε βιοεπεξεργασίας, βιομεταποίησης, Νέε βιομηχανίε θα εξειδικευθούν στα βιοπροϊόντα και σίγουρα θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια εκτελεστική επιτροπή όπως και χρηματοπιστωτική οργανισμοί όπως η ΕΤΕ. Πιστεύω ότι οι περιφέρειες αυτές θα έπρεπε να έχουν ε, κάθε ευκαιρία να μετάσχουν σε αυτήν την ρηξικέλευτη αγορά. Όσο προετοίμαζα την ε, έκθεσή μου, προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να εστιάσω την προσοχή μου στην ε, επίρρωση του ρόλου Ε, των ε, παικτών ε, της αγοράς αλλά και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο φυσικά να στεφθεί με επιτυχία αυτή η νέα κοινή επιχείρηση για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Νομίζω ότι η ορθή προσέγγιση και ο μονόδρομος για την επιτυχία είναι να ξεκινήσουμε από, τα, από κάτω και να ανέβουμε προς τα πάνω ώστε να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή των τοπικών φορέων ε, και κυρίως ε, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί από περιβαλλοντική σκοπιά σε ε, σύσσωμη κοινωνία. Πιστεύω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ακριβώς η ενίσχυση της συνεργασίας των δημοσίων φορέων με την βιομηχανία για την έρευνα. Ο τριπλός έλκας και Πιστεύω ότι με την κοινή επιχείρηση θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να λειτουργήσει αυτή η νέα προσέγγιση. Θα δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση, διότι όλοι οι φορεί τη οικονομική ζωή θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Κατόπιν ασχολήθηκα και με ε, το διανοητικό κεφάλαιο, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δηλαδή ε, αξιοποιήσουμε χρησιμοποιούμε τις, ε, ο, ε, τους όρους που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο, τα όσα ισχύουν για τους γεωργούς. Ξέρετε, μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω, διότι η πρόεδρος μου είπε έχω, ότι έχω περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν και είμαι στη διάθεσή σας ε, για ερωτήσεις. Ε, πρόεδρος, ε, ο κύριος Λάμπρεχ δεν είχε ακουστικά και δεν ξέρει πόσο πολύ τον ευχαριστήσατε για την υποστήριξη και τη βοήθεια του. Το επαναλαμβάνω, Γιάνν Νίλσεν τώρα που είναι σκιώδης για τους σοσιαλιστές θα πάρει το λόγο παρακαλώ.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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση και πιστεύω όντως ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία. Φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όπως πάντα, αλλά πραγματικά εγώ επειδή είμαι στη, ζω στη Βόρεια Σουηδία και εκεί έχουμε το ε, δασικό απόθεμα της Ευρώπης, ε, νιώθω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα και φυσικά ε, τα βιοκαύσιμα που μπορούν να παραχθούν σε μια τέτοια περιοχή ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, τώρα, ε, η διασύνδεση που δημιουργείται με την κοινή επιχείρηση είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει δηλαδή αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που αποφασίζουν να όντως να διασυνδέονται, αλλά ελοχεύει και ένας κίνδυνος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή θα πρέπει να απευθύνουμε σαφή πρόσκληση προς την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δηλαδή μας μιλήσατε για τη Unilever παραδείγματο χάρη. Δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοιους παίκτε να αποφασίζουν αποκλειστικά μόνοι του. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, περιφέρειες ε, που έχουν εκπονήσει εξάλλου και περιφερειακές στρατηγικές για τα βιοκαύσιμα και όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν. Να χρησιμοποιήσουμε επίσης την τεχνογνωσία που έχουμε στην Επιτροπή μας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ούτω ώστε οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων να θεωρηθούν σαν απόσπαστο κομμάτι της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση. Η ίδια η έκανε κάποιες προσθήκες. Ήθελα μόνο να σας προειδοποιήσω ότι ε, διατρέχουμε αυτό τον κίνδυνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να συμμετάσχουν όταν συζητάμε και όταν αποφασίζουμε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Φερνάντες, είναι εδώ, έχετε το λόγο. Από τους πράσινους. Δεν θέλετε να μιλήσετε? Εντάξει. Δεν έχουμε κανένα άλλο μιλητή. Α, ο κ. Φανίστεροι. Ντόψη. Ντόψε. Και στα πολωνικά. Α, αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάω, ε, ότι πολωνικά βέβαια. Κρίμα λέει η πρόεδρος. Στην Επιτροπή Ήτρε θα συζητηθεί το θέμα α, στην ε, Επιτροπή Ήτρα θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις 11 για την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Ειδικά στην Επιτροπή Βιομηχανίας πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν μεγάλοι εταίροι που θέλουν να επενδύσουν ε, πρέπει να υπάρξει μια κοινή ατζέντα και μέσα σε αυτή να υπάρξουν επενδύσεις και κοινή ευθύνη. Έχουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον ακριβή προϋπολογισμό. Και έχουμε 2,8 δισεκατομμυρία ε, επενδύσεων από τη βιομηχανία. Είναι πολύ ε, ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπετε την ε, πλήρη δέσμευση που υπάρχει. Δεν μιλάμε τώρα για μελέτης, μελέτες απλώς, μιλάμε για μια προσπάθεια εφαρμογής των, στις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Θέλω να μιλήσω για την έκθεση της Μπεθ. Υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην διάδοση αυτής τεχνολογίας, όλων των πτυχών αυτής της έκθεσης. Και αν κοιτάξετε στο παρελθόν πώς λειτουργούσαν οι κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, θα βλέπατε ότι υπήρχαν πλούσιες χώρες, Και είχαμε πρωτοβουλίε κυρίως από τα παλιά κράτη-μέλη. Αυτές ήταν μπροστά. Αν μιλάμε για τις περιοχές σύγκληση, για την περιφερειακή πολιτική, τώρα θέλουμε να υπάρξουν κοινέ ε, τεχνολογικές πρωτοβουλίες και στα νέα κράτη-μέλη. Μπορείτε, αν δείτε τη μερίσια διάταξη, να δείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίε παντού. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει, στη Ρουμανία σε πολλές περιφέρειες. Επομένως η διάδοση αυτής της ιδέας και η δημιουργία αυτής της κοινή επιχείρησης, αυτής κοινοπραξίας ε, και η σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η συμμετοχή των επιστημονικών Ινστιτούτων, των ερευνητικών Ινστιτούτων, όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Ο συντονισμός η χρήση των μέσων που έχουμε στο Interreg για να προωθήσουμε τη συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και, και να μην περιοριστούμε μόνο στις περιφέρειες όπου εδρεύουν και οι μεγάλες αυτές εταιρείε. Μιλάμε για μια πολύ πιο ευρεία ατζέντα και συνδέεται πολύ με τις ε, δραστηριότητες της Επιτροπής μας. Πολλές από αυτές τις εταιρείε είναι μπροστάριδες. Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, οι νέες δυνατότητες. Αλλά η εφαρμογή μπορεί να γίνει παντού. Η μετάβαση σε μια, βιομηχανία, σε μια οικονομία βιομηχανιών βιοπροϊόντων έχει τεράστιο δυναμικό. Όχι ίσως... Ε, όχι μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά και σε πολλές περιοχές της υπαίθρου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση. Θα είμαι σε επαφή μαζί σας και θα παρακολουθήσω και την πρόοδο της συζήτησης ε, στην Επιτροπή Ήτρε που θα ξεκινήσει όπως σας είπα στις 11. Ευχαριστώ Λαμπέ. Ο κύριος Φερχάχτερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει, παρακαλώ αν θέλει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι στη Γενική Διεθνή Έρευνα και Καινοτομίας. Ε, είμαι ευγνώμων για, την, ε, για τα θαυμάσια και θερμά σχόλια της εισηγήτριας. Ε, μας υποστηρίζουν, θαυμάσια η έκθεση, πλήρης, μας βοηθάει. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εντάξουμε και την περιφερειακή διάσταση. Αν θέλουμε ε, ευρωπαϊκές τέτοιες βιομηχανίες βιοπροϊόντων, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία ε, περιφερειακή προσέγγιση. Θα πρέπει να την εντάξουμε πλήρως στην πολιτική μας και να την ενισχύσουμε. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνουμε, όταν κάνουμε την πρόταση για, συμβούλιο, για κανονισμό του Συμβουλίου, ε, εκεί θα εντάξουμε και μέτρα περιφερειακής πολιτικής. Ένα σχόλιο που έκανε ο κύριος Φανίστελ Ρόι. ο κύριος Νίλσεν, συγγνώμη. Είναι σημαντικό μια τέτοια πρωτοβουλία να είναι ανοιχτή, διαφανής σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Να μην είναι ένα κλειστό κλαμπ, δηλαδή, αυτό που θα κάνει αυτές τις δουλειές. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει ευρεία συμμετοχή, εμπλοκή όλων των φορέων και των περιφερειακών αρχών. Ειδικά οι περιφέρειες στη φάση της ανάπτυξης της πρωτοβουλίας θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο. Ε, πρόκειται για προγράμματα έρευνας και καινοτομία λοιπόν, τα οποία προτείνονται. Η θαυμάσια έρευνα και η θαυμάσια καινοτομία δεν αρκεί αν δεν αναπτυχθούν συνεχεία αυτά τα προϊόντα, αν δεν μπουν στην αγορά, αν δεν φτάσουν οι υπηρεσίες αυτές στον καταναλωτή. Και αυτές οι πρωτοβουλίες θα δημιουργήσουν ε, ευκαιρίες για τις περιφέρειες ε, των κρατών μελών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τελευταίες παρατηρήσεις από την εισηγήτρια. Θέλετε. Ναι, θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά τους. Χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε για το ότι είναι σημαντικό και ότι είναι πολύ σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξουν οι περιφέρειες ε, και ότι πρέπει να τις εντάξουμε ενεργά, ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια να, να τελεσφορήσει. Πιστεύω ότι αν δημιουργηθεί αυτή η κοινή επιχείρηση, θα ε, έχουμε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολυτεχνία κυρίως ερευνητικά κέντρα κτλ. Όλοι αυτοί θα μπουν έτσι πολύ θερμά σε αυτή την πρωτοβουλία, θα ενταχθούν. Ευχαριστώ. Η Ήτρε θα εγκρίνει αυτή την έκθεση σε 9 Ιανουαρίου. Οπότε η μόνη μας επιλογή είναι να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο. Γι' αυτό προθεσμία υποβολή τροπολογιών 28 Νοεμβρίου το μεσημέρι, πολύ βέβαια περιορισμένη. Ωραία. Να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερής διάταξης. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Σιλάγκη ε, θα αντικαταστήσει τον κύριο Γκοτμάνης για τις στατιστικές ε, σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ευχαριστώ. Από πλευράς του Ήβαρς Γκοτμάνης. Ζητάω συγγνώμη που δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ε, συνεδρίασή μας. Θα παρουσιάσω λοιπόν τη γνωμοδότησή του για την ποιότητα των στατιστικών που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η πρόταση της Επιτροπής έχει εκπονηθεί για να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Απασχόληση και Ανάπτυξη. Η Επιτροπή ε, παράλληλα με τα υπάρχοντα μέτρα δημιουργεί, έχει θέσει κανόνες για την ε, έγκαιρη ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των ανισορροπιών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο συγητής τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά ε, διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μαζί με το γεωργικό και το αλληλευτικό ταμείο είναι ένα σημαντικό τμήμα των δημοσίων επενδύσεων πολλών κρατών μελών και περιφερειών. Και η αναστολή του θα μπορούσε να αυξήσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αν ανασταλεί η χρήση κάποιων ταμείων, η χορήγηση ε, πιστώσεων από κάποια ταμεία, δεν θα πρέπει να είναι παρά μόνο το τελευταίο μέτρο που θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από σε βάθος ανάλυση της μείωσης του ΑΕΠ, ε, της ε, φτώχειας και της ανεργίας. Είναι σημαντικό να έχουμε υψηλού επίπεδου και έγκαιρα στατιστικές. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τονίζει ότι για να υπάρχει συνεπής εφαρμογή της διαδικασίας ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλού επίπεδου στατιστικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Υποστηρίζει λοιπόν ο συγητής την πρόταση τη Επιτροπής ότι πρέπει να είναι ανοιχτό ο κατάλογος των δικτών που θα πρέπει να αναλύονται και προτείνει ακριβώς αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ουκατσέσκα, Σκιώδης του ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι πρόκειται για πάρα πολύ εύστοχες ε, τροπολογίες ε, χάρη στατιστικές ε, μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση, θα έχουμε μια ταχύτερη αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. είναι θεμελιώδους ε, σημασίας ε, να συνεχίσουμε την εποπτεία και να έχουμε διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την ε, ΜΥΠ, τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, ανά πάσα στιγμή. Είναι λοιπόν Προφανή η σημασία των στατιστικών στοιχείων, διότι μόνο με τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να διασκεδάσουμε οποιασδήποτε ανησυχίες υπάρχουν. Είναι σημαντικό να δούμε ποια ορολογία θα χρησιμοποιείται, ποιες μέθοδοι θα ε, χρησιμοποιηθούν για να εκπονηθούν οι δείκτες αρχικά και ε, μεταγενέστερα τα στατιστικά στοιχεία για τη συνεργασία με τα εθνικά ε, στατιστικά Ινστιτούτα θα πρέπει να μεριμνήσουμε επίσης ούτω ώστε να έχουμε μια διασυνοριακή προσέγγιση αλλά και ε, να τονίσουμε την σημασία του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου διότι ε, η ανάπτυξη και η πορεία της οικονομίας δεν μπορεί να κρίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο ε, αλλά θα πρέπει ε, να κατέβουμε και στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Συμφωνώ λοιπόν με όλες τις προτάσεις που ακούσαμε και τις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Νίκος Χρυσόγελος ε, για τους πράσινους. Ε, ε, είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα στατιστικών δεδομένων και φυσικά σωστούς δείκτες, αλλά και σωστές εκθέσεις και επίσης ε, μια συνολική εικόνα τι γίνεται σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ε, πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε σωστά και τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη και δεν πρέπει ε, να, ε, πρέπει μάλλον να έχουμε ένα ανοιχτό κατάλογο των δικτών και όμως πρέπει να ξανασυζητήσουμε πώς οι δείκτες ε, οι μακροοικονομικοί αντιπροσωπεύουν ε, και αλληλοσχετίζονται επίσης με θέματα κοινωνικής συνοχής, ανισοτήτων, περιβάλλοντος, εκπαίδευση κλπ. Δηλαδή πολλές φορές οι δείκτες δεν περιγράφουν τη σωστή πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να στήσουμε περισσότερο. Δηλαδή παρότι μιλάμε για μακροοικονομικούς δείκτες, αυτοί πρέπει να ελοσχετίζονται και με την υπόλοιπη κατάσταση οικονομίας γιατί πολλές φορές τα νούμερα παραπλανούν. Δηλαδή αν πετύχουμε ε, μια εξυγίανση ε, των ελλημάτων ή του χρέους πρέπει να ξέρουμε και πώς έχει γίνει αυτό, τι αποτελέσματα είχε πάνω σε άλλους σε άλλες ε, καταστάσεις όπως είναι η κοινωνική συνοχή ή το περιβάλλον. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι μια ζήτηση που φαντάζομαι θα κρατήσει αρκετό καιρό. Με αυτή την έννοια είναι σωστό όταν συμφωνήσουμε στους κανόνες, τα κράτη-μέλη να τηρούν τους κανόνες και να υπάρχουν και κυρώσεις. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση, αν το ύψος των κυρώσεων είναι αυτό που περιλαμβάνεται στην έκθεση ή πρέπει να είναι μικρότερο, ή μας συλλογική να είναι μικρότερο. Αλλά εδώ υπάρχουν και δύο θέματα. Ε, ποιο τελικά πληρώνει τι κυρώσει, γιατί πολλέ φορέ αυτό τιμωρεί την κοινωνία και όχι την κυβέρνηση ή τους, τις στατιστικές αρχές που ε, έχουν κάνει την κακή έκθεση, την, ε, την αλλίωση των, ε, στοιχείων. Και το δεύτερο, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το βάρος στην απόφαση, το, η απόφαση να παίρνεται κυρίως από το Ευρωκοινοβούλιο και όχι τόσο από το Συμβούλιο. Έχουμε δει πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ε, θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει να είναι σαφές και στην έκθεση ότι έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι κυρώσεις γιατί δεν παρέχονται σωστά στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις. Από την άλλη μεριά είμαστε πλήρως αντίθετοι να συνδέεται αυτό με επιβολές κυρώσεων στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στι περιφέρειε, όπω είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε να μην συζητήσουμε στην Ολομέλεια, για το θέμα των κυρώσεων σε περίπτωση μη επίτευξη μακροοικονομικών στόχων. Δηλαδή, επειδή μένει ανοιχτό το θέμα εδώ και απλώ είναι πιο ήπιε οι διατυπώσει στην έκθεση, εμεί δεν θα θέλαμε να ψηφιστεί μέσα στην έκθεση οποιαδήποτε αναφορά σε κυρώσει εάν δεν επιτυγχάνονται οι μακροοικονομικοί στόχοι όχι αν δεν είναι καλή ποιότητα των δικτών ή των εκθέσεων. Thank you. I, don't see any other... Δεν, μιλάει δεν θέλει άλλο στο λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, αλλά έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν και στον εκπρόσωπο της Eurostat που θα πάρει το λόγο σε λίγο. Το ερώτημά μου είναι, αν έχουμε ένα επαρκώς αναπτυγμένο σύστημα για να μετρήσει και τις ε, επιπτώσεις των μακροοικονομικών ανισορροπιών, δηλαδή τις επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Ο εκπρόσωπος της Eurostat θα ήθελα να μου απαντήσει παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως να απαντήσω αμέσως ε, στην ερώτησή σας. Όντως, ε, ε, ξέρετε, έχουμε ένα, ένα πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων ε, και άλλους συμπληρωματικού δείκτες. Δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013. Αν δεν απατώμε, υπάρχουν 8 δείκτες που σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα. Οπότε ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλήρες ε, σετ ε, δεδομένων που θα, υποστηρίζουν, θα λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς την οικονομική μας ε, ανάλυση και ως προς τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, αλλά και ως προς τις πιθανές επιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα να προσθέσω ε, πως ε, είναι προφανές ότι έχουμε εξετάσει το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής σας και πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που εμπεριέχει είναι ένα καλό εφαλτήριο για τις μελλοντικέ μας συζητήσει. Τα στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας για να υποστηριχθεί η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι, είναι κάτι απαραίτητο για μας. Ως εκ τούτου ε, καταθέτουμε αυτή την πρόταση ώστε να θεσπίσουμε ένα ισχυρό ε, πλαίσιο ε, για την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων ώστε να βασιζόμαστε σε αδιαμφισβήτητα γεγονότα και δεδομένα για την περαιτέρω οικονομική ανάλυση. Ε, από αυτή τη σκοπιά υποστηρίζουμε την δική σας πρόταση για ποιοτικά ε, στοιχεία ε, στήριξης της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το σχέδιο επίσης ε, αναφέρεται ότι η ενδελεχής ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνεκτιμά και τις συγκυρίες που ισχύουν σε κάθε συγκεκριμένη χώρα, κυρίως ως προς τα κοινωνικά ζητήματα, την απασχόληση, την ανεργία, την οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη, την ε, εξέλιξη του ΑΕΠ. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο και αυτό θα πράξουμε ούτως ή άλλως. Ως προς τις κυρώσεις, οι κυρώσεις έχουν ως στόχο να πατάξουν ε, αποκλειστικά και μόνο την αλλίωση των στατιστικών στοιχείων που θεωρούμε απαράδεκτη. Ε, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα πρέπει να αποτρέπει ονδήποτε από την αλλίωση των στατιστικών στοιχείων και αυτός είναι ο στόχος και ε, η φύση των κυρώσεων. Επαναλαμβάνω και τονίζω ότι στοχεύουμε μόνο την ε, αλλίωση η οποία έχει γίνει εσκεμένα ή προέρχεται από σοβαρή αμέλεια. Αυτά, Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό το στάδιο. σε ευχαριστώ. Ο Νίκος, από ό,τι κατάλαβα, θέλει να δευτερολογήσει, να αναφερθεί σε αυτά που είπατε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα ε, ξέρουμε ότι πολλές φορές αλλάζουν τα στατιστικά δεδομένα και στην αρχή της κρίσης όσον αφορά την Ελλάδα υπήρξε διαφοροποίηση ως προς το τι περιλαμβάνεται τα στατιστικά στοιχεία για μακροοικονομικά θέματα, π.χ. το θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα ή άλλα. Ε, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πάντα μια σταθερή, ε, μια, μια εντελώς ξεκάθαρη ε, απόφαση ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στους δείκτες της εκθέσης. Αλλά έχω την εντύπωση μια δεύτερη ερώτηση ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των στατιστικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις μακροοικονομικές εκτιμήσεις για την Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Τουλάχιστον έχω διαβάσει κάποια άρθρα γι' αυτό. Ε, το δεύτερο είναι σε σχέση με αυτό που είπατε αρχικά. Κοινωνικοί δείκτες σήμερα από την Τρόικα δεν λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή όλη η συζήτηση για την ε, δημοσιονομική εξυγίανση δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια κατάρρευση που υπάρχει σε κοινωνικό και σε παραγωγικό επίπεδο. Είπατε ότι υπάρχουν 8 δείκτες στους οποίους ε, συνυπολογίζουμε, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην πολιτική για τα δημοσιονομικά. Άρα οι δείκτες είναι εκεί, μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά πώς επηρεάζει τις πολιτικές για τα δημοσιονομικά. Δηλαδή πώς συνδέεται αυτό στην πράξη με πολιτικές δημοσιονομικές προσαρμογής. Ε, νομίζω, Νίκο, προ την ΕΚΦΙΝ και όχι προ την Eurostat έπρεπε να απευθύνει την ερώτησή σου, αλλά ευπρόσδεκτη και απάντηση. Παρόλα αυτά, ο Όλτζι Βλάσακ θέλει να δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα αυτή τη συζήτηση. Και νομίζω ότι ένα μήνυμα είναι αυτό που περνάει τελικά. Ότι χρειαζόμαστε καλές στατιστικές για να λειτουργεί ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχουν προβλήματα με αυτό, τουλάχιστον να αναγκαστούν οι διάφορες αρχές να ενοποιήσουν τη μεθοδολογία τους, να την να πλησιάσουν μία την άλλη. Άρα σωστή είναι η έκθεση. Λοιπόν, τώρα ο συνάδελφος από την Eurostat και μετά ο εισηγητής. Χωρίς μικρόφωνο. Το ερώτημα νομίζω ότι απευθύνεται περισσότερο τη συνέχεια που θα δοθεί στις ε, δημοσιονομικές πολιτικές. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι αρμοδιότητα της ΕΚΦΗΝ. Τώρα, σε σχέση με αυτή την πρόταση, έχω να πω το εξή. Υπάρχει ο μηχανισμός ε, προειδοποίησης, η έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν τον Νοέμβριο. Κάναμε μία ανάλυση για κάθε χώρα και λάβαμε υπόψη όχι μόνο καθαρά μακροοικονομικούς δείχτες, αλλά και μια σειρά από άλλους κοινωνικούς δείκτες. Αυτό είναι ο στόχος της, των εκθέσεων αυτών και προσπαθούμε να δώσουμε στατιστικά στοιχεία που να καλύπτουν και άλλες πτυχές, όχι μόνο τις μακροοικονομικές αλλά και τις κοινωνικές. Το θέμα για την Τρόικα και τις μακροοικονομικές πολιτικές όμως νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσει η Τρόικα. Ευχαριστώ. Τελικά σχόλια τον εισηγητή παρακαλώ. Από το Σιλάγκη. Προέρχονται. Ε, ε, μιλάω εξ ονόματος του εισηγητή, τον κύριο Γκοντμάνης. Πιστεύω ότι θα προτείνει συμβαστικές τροπολογίες μετά από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, ούτως ώστε ε, να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες αυτές και από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα υιοθετηθεί στις 13 Φεβρουαρίου από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες. Επομένως, να έχουμε προθεσμία μέχρι 2 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε λοιπόν μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους και τη Eurostat. Και τώρα πάμε στο σημείο 6 της ε, ημερήσιας διάταξης. Ζέλερ. Ο κύριος Ζέλερ είναι μαζί μας, η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Μάρτιο η Επιτροπή δημοσίευσε μια πράσινη βίβλο όπου έθετε αρκετά πολλά ερωτήματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των νέων κανόνων για τη ρύθμιση και την σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις επιπτώσεις ε, που θα είχαν όλα αυτά στη δημιουργία έργων υποδομής και στις ε, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συζητιέται από την ΕΚΟΝ, αλλά νομίζω ότι και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιφερειακής ε, δραστηριότητας ε, επηρεάζονται και αυτές. Διότι αν υπάρχουν προγράμματα έχουν μία ε, σίγουρη μακροπρόθεσμη βάση λειτουργίας. Και γι' αυτό θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα αυτό. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κίνδυνος δυσχεριών μέσω αυτών των νέων κανόνων αλλά και των μέτρων για την εξυγίαση και σταθεροποίηση των τραπεζών, δηλαδή το ποσοστό ιδίου κεφαλαίου που απαιτείται από τις τράπεζες, αλλά και η πιο αυστηρή αποτίμηση του κινδύνου των προγραμμάτων. Οπότε υπάρχει κίνδυνος ε, για τα πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα. τα προγράμματα δηλαδή που χρειάζονται πολλά χρόνια για να εκτελεστούν πλήρως. Μπορεί να φυγούν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μία σφαιρική εικόνα. Να δούμε δηλαδή τι έχουμε. Εμείς ε, τα διαθροτικά ταμεία τα θεωρούμε ε, τμήμα των δημοσίων επενδύσεων, αλλά υπάρχουν και εθνικές δημόσιες επενδύσεις, υπάρχουν και δυνατότητες εθνικής χρηματοδότησης από τις τράπεζες και άλλα εθνικά χρηματοδοτικά μέσα αρμοδιότητας ε, μεμονωμένων κρατών μελών. Και υπάρχει και το θέμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης, που θα έπρεπε και αυτή να βοηθήσει μαζί με τις δημόσιες τράπεζες και υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ε, ορισμένα εκ των οποίων έχουμε ήδη αποφασίσει και των οποίων αποτελεσματικότητα και αυτή θα μπορούσε να επηρεαστεί. Είδαμε λοιπόν ότι επειδή είμαστε σε περίοδο κρίσης, η οποία ακόμη ε, δεν έχει πλήρως υπερνικηθεί, η κρίση λοιπόν έχει τρομερές επιπτώσεις για τις μικρομεσαίες γιατί δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση. Και στα κράτη-μέλη όπου δεν υπήρχαν για τις επιχειρήσεις ήδη υπογεγραμμένα μακροχρόνια συμβόλαια, δημιουργήθηκαν πολλές δυσχέρειες ακριβώς επειδή υπήρξε και μεγάλη διακύμανση των επιτοκίων. Και επειδή διεκόπη απλά και μόνο η δημόσια χρηματοδότηση κάποιων μακροπρόθεσμων μεγάλης έκτασης προγραμμάτων και έπρεπε να εξευρεθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό έκανα προσπάθεια, σύντομα βέβαια, να διατυπώσω μια γνωμοδότηση που περιέχει 8 σημεία πώς θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε στο μέλλον να διασφαλίσουμε τα μακροπρόθεσμα προγράμματα και μέσω δημοσίων επενδύσεων αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι όπως ξέρετε η ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομιών. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι φυσικά ο περιορισμός της χρηματοδότησης σε κάποιες ε, χώρες που ε, πλήττονται από την κρίση έχει ως συνέπεια η δημόσια χρηματοδότηση να έχει περιοριστεί πολύ ή απλώς να έχει διακοπή. Γι' αυτό χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα χρηματοδότησης για να αντικαταστήσει αυτές τις ελλείψεις. Κάτα τις μελέτες μας διαπιστώσαμε Ας δούμε για παράδειγμα το γερμανικό παράδειγμα. Οι μικρομεσαίες ε, ε, χρηματοδοτικές πηγές, για μας για παράδειγμα τα ταμιευτήρια στη Γερμανία, σε συνθήκες κρίσης ήταν οι πιο σταθερές εναπομένουσες πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό προτείνουμε στην Κομισιόν να προσέξει ιδιαίτερα αυτές τις πηγές ε, χρηματοδότησης, ούτως ώστε οι συνεταιριστικές, οι κοινωνικές ε, τράπεζες, δηλαδή οι τράπεζες σε, δημόσιο, σε δημοτικό συγγνώμη, ή περιφερειακό επίπεδο, αυτές μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ να επιβιώσει το σύστημα χρηματοδότησης. Να μην τους επιβάλλουμε δηλαδή τέτοιες υποχρεώσεις που τελικά να μην μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει δισεκατομμύρια μέσα από διάφορα μέσα για να διασφαλιστούν κάποιες επενδύσεις και δεν αξιοποιήθηκαν. Οπότε θέτω το ερώτημα. Δεν ήταν γνωστά αυτά τα μέσα ή ήταν ε, υπερβολικές ε, οι ανάγκες των προγραμμάτων δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε όλες και ποικίλε, όλες τις ποικίλε δυνατότητες της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας, μια που οι κλασικές πηγές έχουν στερέψει, για να συνεχιστούν τα μακροπρόθεσμα προγράμματα. Δυστυχώς διαπιστώσαμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει δισεκατομμύρια στις ιδιωτικές τράπεζες για να προκαλέσει επενδύσεις. Αλλά δυστυχώς αυτά τα δισεκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν για να εξηγιάνουν τις τράπεζες. Δεν μεταφράστηκαν σε επενδύσεις, τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε δημιουργήθηκαν μια σειρά προβλήματα. που κατά την άποψη της Περιφερειακής Επιτροπής από τη δική μας οπτική γωνία θα έπρεπε να αναφερθούν. Προσπάθησα να το εκφράσω στο κείμενο της γνωμοδότησης και νομίζω ότι μέσω των τροπολογιών των συναδέλφων μπορούμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο ούτως ώστε να το αποστείλουμε στην ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Μόιτσα Κλέβερ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ΕΚΟΝ είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και ασχολήθηκε αυτή τη βδομάδα με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να συμπεριληφθούν και οι δικές μας απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Ευχαριστώ την εισηγητή για τη θαυμάσια έκθεση. Το σχέδιο γνωμοδότησης μας υποβλήθηκε εγκαίρως. Έχουμε πολύ χρόνο λοιπόν για τη σύνταξη της νομοδότησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και είμαι πεπισμένη ότι η πολιτική συνοχής θα παίξει σημαντικό ρόλο, για να μην πω τον πιο σημαντικό ρόλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το, τα ταμεία συνοχής είναι τα ταμεία τα οποία οδηγούν σε καλύτερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη, σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, σε μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε το ρόλο των τραπεζών πριν και μετά την κρίση. Η δανειακή τους, το δανειακό τους δυναμικό δεν επαρκεί και σήμερα όμως με την κρίση δεν μειώνουν τις προϋποθέσεις για δάνεια. Αυτά τα δάνεια όμως είναι απαραίτητα σε ιδιώτες, σε νοικοκυριά κτλ. Η τραπεζική κρίση είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ πηγές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η μέσα καινοτόμας χρηματοδότησης θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Μιλάμε για αυτά τα πράγματα όχι μόνο σε αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά τα εντάξαμε και, στο, και στη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Στο 7ο πάντως, για το 7ο πολιετές πρόγραμμα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αυτά τα, αυτοί οι μηχανισμοί, αυτά τα μέσα θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της γρήγορης και διαφανούς εφαρμογής νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε και ένα πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Και επίσης οι σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού εδώ έχουν ε, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης ε, πάρα πολύ διαφάνεια για τη χρήση των ε, άτυπων χρηματοδοτικών μέσων ε, και να ξέρουν τα κράτη-μέλη πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και πού να τα βρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον, για αυτά τα άτυπα μέσα χρηματοδότησης. Ε, τα μη επίσημα, ας πούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τέλος τον εισηγητή για τη θαυμάσια γνωμοδότηση και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Από τους πράσινους ο Νίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα ουσιαστικό πρόβλημα, δηλαδή τη χρηματοδότηση μακροχρόνια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, και αυτό είναι σημαντικό όχι αφηρημένα, αλλά γιατί πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες, να στηριχθεί η κοινωνική ένταξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, και να πετύχουμε στόχους οποίους έχουμε θέσει. Δηλαδή οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ή στόχοι για ε, κοινωνική συνοχή, αυτοί δεν θα επιτευχθούν ποτέ αν δεν υπάρχει πραγματικά μακροχρόνια χρηματοδότηση οικονομίας, αν κάθε κρίση διακόπτει τη χρηματοδότηση. Οπότε αυτό θα ζητάμε ωραία για πολιτικές, αλλά δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα σήμερα, ότι η κρίση και η ύφεση έχουν αυξήσει τις ανισότητες. Μπορεί να προσπαθούσαμε πολλά χρόνια να μειώσουμε τις ανισότητες. Είναι η πρώτη φορά που τώρα αυξάνονται οι ανισότητες και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πώς θα αλλάξουμε τις στρατηγικές μας. Αυξάνονται οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, αλλά και στο εσωτερικό των περιφερειών. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε δείκτες ΑΕ που δείχνουν ότι μια περιφέρεια είναι αναπτυγμένη αλλά δημιουργούνται πολλές εστίες μέσα στις περιφέρειες που έχουν μεγάλα προβλήματα είτε λόγω αυξημένης ενεργείας είτε ε, απουσίας κοινωνικής συνοχής. Απ' την άλλη, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ενώ χρειαζόμασταν περισσότερους πόρους δημόσιους, για πρώτη φορά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι μειωμένος. Έχουμε παράλληλα μείωση των διαθέσιμων εθνικών πόρων σε πολλές περιοχές, αλλά και των ιδιωτικών πόρων, τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχουν χρήματα ε, στην οικονομία παγκοσμίω, αλλά δεν σημαίνει ότι κατευθύνονται εκεί που υπάρχει ανάγκη, δηλαδή στις περιφέρειες και στις ε, κοινωνίες για να μειώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, και το επιπλέον πρόβλημα είναι ότι έχουμε και μεγάλο πρόβλημα στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Και γιατί πολλές τράπεζες είναι εκτεθειμένες αλλά και επειδή έχει αυξηθεί το ρίσκο και οι τράπεζες πλέον ακόμα και υγιείς επενδύσεις και υγιείς οικονομικές δραστηριότητες δεν χρηματοδοτούνται εύκολα από τις τράπεζες. Ξέρω στην Ελλάδα ότι το 80% των αιτήσεων, ακόμα και για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τράπεζες απορρίπτουν λόγω των γενικότερων δυσκολιών που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα τη στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση, σχεδόν όλες οι πηγές χρηματοδότησης έχουν κλείσει. Καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να εξηγιάνουμε, να αλλάξουμε το τραπεζικό σύστημα, να είναι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και να εκπληρώνει το ρόλο του, τον κύριο ρόλο του που είναι η χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας αυτό πρέπει να επανέλθει και γι' αυτό η, τραπεζική εποπτεία, η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και η εξυγίανσή τους είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να πληρώνει γι' αυτό συνεχώς η κοινωνία. Αλλά δεν μπορεί συνέχεια να πληρώνουμε τεράστιο κόστος στις τράπεζες για εξυγίανση αλλά αυτοί οι πόροι να μένουν στις τράπεζες. Το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης διαθέτει 50-60 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ίσως χρειαστούν και περισσότερα, αλλά δεν φτάνει σχεδόν τίποτα από αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν στραγγίξει. Ούτε εξαγωγές μπορούν να κάνουν, ούτε τίποτα από τη στιγμή που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί τις τράπεζες, δίνει κεφάλαια στις τράπεζες, δεν χρηματοδοτεί όμως τα κράτη-μέλη της περιφέρειας. Πώς θα φτάσουν τα χρήματα στην πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν, πρώτον, πρέπει να εξηγιάνουμε το τραπεζικό σύστημα και οι πόροι που διατίθενται να φτάνουν στην πραγματική αγορά. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η τεράστια απουσία ρευστότητα στην οικονομία. Το δεύτερο που σωστά επισημαίνει η έκθεση είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Ε, παράδειγμα, οι συνεταιριστικέ τράπεζε στι περισσότερε χώρε είναι σε υγιή βάση, έχουν εκτεθεί πολύ λιγότερο. Άρα πρέπει πράγματι, όπως είπε και ο συγητή οι κανόνες εποπτείας να λάβουν υπόψη ότι δεν έχουν εκτεθεί, δεν έχουν προκαλέσει τα ίδια προβλήματα με το συστημικό τραπεζικό σύστημα, άρα οι κανόνες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην πραγματική εικόνα των συνεταιριστικών τραπεζών και είναι ένα κατάλληλο εργαλείο γιατί οι περισσότεροι πόροι τους πάνε στην τοπική οικονομία και στις επιχειρήσεις και στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη οι συστημικές τράπεζες πολύ δύσκολα δίνουν χρήματα στο συνεταιριστικό τομέα και στην κοινωνική οικονομία, τη στιγμή που και δικές μας εκθέσεις έχουν επισημάνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι τεράστιος ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να δημιουργηθούν θέσεις εργασία και ε, να μειωθεί η ανισότητα. Άρα λοιπόν σίγουρα πρέπει να δούμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις συνεταιριστικές τράπεζες Πρέπει να δει και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη κατάλληλα εργαλεία για ομόλογα έργου και στο περιφερειακό και στο εθνικό επίπεδο. Το μοντέλο που υπάρχει ακόμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι για μεγάλα project που δεν είναι εύκολο να μπουν οι περιφέρειες και από την άλλη μεριά οι περιφέρειες δεν έχουν ένα ευέλικτο σύστημα για ομόλογα έργου και κυρίως για πράσινα ομόλογα όταν θέλουμε να κάνουμε επενδύσει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπω λέγαμε στην προηγούμενη συζήτηση, παράδειγμα για ευφυή δίκτυα. Άρα λοιπόν πρέπει το σύστημα να εξειδικευθεί και να μπορέσουμε να έχουμε αξιόπιστα μοντέλα εναλλακτική χρηματοδότηση, αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι μόνο μεγάλα project 50 εκατομμυρίων και πάνω. Και το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα χρηματοδοτήσει χώρε που έχουν προγράμματα δημοσιονομική προσαρμογή και δεν έχουν πετύχει του δημοσιονομικού στόχου, αλλά αν εφαρμοστεί και η, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αυτό θα το κάνουν επίση και οι ιδιωτικέ τράπεζε ή άλλε τράπεζε. Δηλαδή, ο κίνδυνο είναι οι χώρε που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά και κοινωνικά, λόγω του καθεστώτος της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, να μην μπορούν να πάρουν χρηματοδοτήσεις και από αναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης. Επομένως, πώς θα στηρίξουν τη χρηματοδότηση ή προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Και λέω μερικά πρέπει επίσης να βρεθούν τρόποι σε όλες τις χώρες για τις λεγόμενες μικροπιστώσεις. Είναι μια δικασία που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους και για φορείς κοινωνικής οικονομίας που χρειάζονται μικρά κεφάλαια τα οποία δεν βρίσκουν. Εύκολα ή σχετικά εύκολα μπορεί να βρει κάποιο κεφάλαια. Είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση και θέλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά πολύ δύσκολα βρίσκει χρήματα κάποιο που είναι μικρό, ένα νέο άνεργο που χρειάζεται 2, 3, 5.000 ευρώ για να ξεκινήσει κάτι, γιατί αν πάει σε μια τράπεζα δεν θα πάρει εύκολα ή θα χρειαστεί πολύ μεγάλε εγγυήσει κατοικία και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλά κάποιος με 3 ή 5.000 ευρώ μπορεί να ξεκινήσει πραγματικά βιώσιμες δραστηριότητες οικονομικές. Ε, πρέπει επίσης να προβλέψουμε αυτό που το Κοινοβούλιο έχει αφασίσει ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιριστικέ επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, θα είναι επίσης δικαιούχοι στα διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από, το ευρωπαϊκό, από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Σα αναφέρω ότι τουλάχιστον στη χώρα μου και σε ορισμένε άλλε που ξέρω, είναι μειονέκτημα αν, έχεις, αν είσαι σε μια συνεταιριστική επιχείρηση και είναι λόγος αποκλεισμού από προγράμματα. Ξέρω πολύ καλά αιτήσει που έχουν γίνει σε διάφορα προγράμματα και αποκλείστηκαν για μόνο λόγο ότι ήταν συνεταιριστικέ και κοινωνικέ επιχειρήσει. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν διακρίσει τέτοιου είδου στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει πάρα πολύ. Νομίζω στην έκθεση θα πρέπει να επισημανθεί πάρα πολύ και θα καταθέσουν και σχετικές τροπολογίες ότι πρέπει να έρθουν όλα τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών. Ε, αυτά ήθελα και θα καταθέσουμε προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης ε, της έκθεσης που είναι ε, σημαντική και ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ, Ιώσεφ Μάτουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, όπως και οι προλαλήσαντες, να τονίσω και πάλι τα όσα έχουμε ήδη ακούσει Όντως είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλους αλλά κυρίως για τα νέα σε εισαγωγικά κράτη-μέλη. Γιατί το λέω αυτό. Διατρέχοντας το σχέδιο έκθεσης για την 7η και 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική συνοχής, που είναι το επόμενο σημείο που θα συζητηθεί σήμερα, βλέπουμε πως η χρηματοοικονομική κρίση ανέστρεψε ε, την ε, διαδικασία σύγκλησης, διεύρυνε το χάσμα που χωρίζει τις επιμέρους περιφέρειες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πλέον αρνητικός αντίκτυπος σημειώθηκε στις ασθενέστερες περιφέρειες ε, και περιοχές ε, της Ένωσης. Στην Ρουμανία, στη χώρα μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για άλλες γειτονικές χώρες, αυτό που συνέβη είναι ότι σώσαμε τις ε, τράπεζες από την κρίση. Όμως οι τράπεζες από πλευράς τους κάνουν αυτό που τους αναλογεί για να σώσουν τη χώρα από την κρίση. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα που θα είναι εγκαίρως προγραμματισμένα μπορούν να μας βοηθήσουν. Ε, αλλά στη Ρουμανία και σε άλλα κράτη-μέλη ε, έχει εμπλακή κατάσταση διότι ε, δεν είναι πλέον διαθέσιμη απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ε, πρόκειται για προγράμματα δημόσιας διοίκησης, προγράμματα για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιέργως πώς ε, δίνονταν πάρα πολύ εύκολα τα δάνεια πριν από την κρίση. Ταυτόχρονα οι χώρες μας τώρα που κάνουν σοβαρές προσπάθειες δεν έχουν διαθέσιμη χρηματοδότηση. Στη Ρουμανία τουλάχιστον ε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη και πόδινη έλλειψη χρηματοδότησης και έχουν εγκαταλειφθεί και καταρρεύσει προγράμματα ακριβώς ε, λήψη χρηματοδότησης. Ο κύριος ε, Τσέλερ μας μίλησε για τις συνεταιριστικές τράπεζες και μοντέλα στήριξης από πλευράς τραπεζών. Όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, δεν θέλω να με παρανοήσετε. Και δεν ε, εξετάζω εδώ την κατάσταση στη Ρουμανία και μόνο. Δεν ε, είναι ιδιαίτερα ιδιάζουσα η κατάσταση στη Ρουμανία. Ε, πάνω από το 90% των τραπεζών έχουν αποκρατικοποιηθεί στη Ρουμανία και λειτουργούν δυνάμει των διαδικασιών που έχουν θεσπίσει οι τράπεζες που έχουν ιδρύσει τις τράπεζες στη Ρουμανία, δηλαδή οι τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης. Ε, ως εκ τούτου υπάρχει προβλεψιμότητα και μέσω μακροπρόθεσμα έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Καλωσορίζω επίσης τις προτάσεις ε, του κυρίου Τσέλερ. Πιστεύω θα μπορέσουμε να τις ε, ενισχύσουμε και να ακουστεί και η δική μας ε, φωνή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει κανένας που να θέλει το λόγο. Όχι, έτσι δεν είναι. Όλτζι Μπλάσεκ, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσέλε και να διευκρινίσω και εγώ ότι χρειαζόμαστε αυτή την έκθεση και κυρίως μια μελλοντική προοπτική. Λυπάμαι που δεν εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι γνωρίζουμε όλοι ε, τα προβλήματα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011 είχε εγκριθεί ένα σχέδιο που στόχο είχε να ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Ήθελα να ρωτήσω του εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιε πρωτοβουλίε τελικά ανελήφθησαν βάσει αυτού του σχεδίου και ποιε έπονται. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πληρέστερη εικόνα για να ολοκληρώσουμε την έκθεση του κ. Τσέλα. Δυστυχώ όμω δεν εκπροσωπείται η Επιτροπή σήμερα, πρόεδρο. Έχουμε του συναδέλφου από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρίτζιο, αλλά αυτή η έκθεση είναι αρμοδιότητα τη ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εσωτερική αγορά αν, κατα... αν κατάλαβα καλά, ε, από το χρηματοπιστωτικό τμήμα. Ε, δυστυχώς στις 28 ήδη λίγη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες, διότι πρέπει να εγκριθεί η έκθεση τον Δεκέμβρη, γιατί η Οίκον θα την εγκρίνει τον Ιανουάριο. Δεν έχουμε χρόνο και πραγματικά θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλια της Επιτροπής. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να γίνει και αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να αποφασίσουμε για τις τροπολογίες. Αύριο το μεσημέρι ναι, Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη, θα σας δώσω, θα σας δώσω το, το λόγο μόλις τελειώσω την πρότασή μου. Όπως είπε και ο συνάδελφος έχει σταλεί η έκθεση ε, στους σκιώδεις και στους συμβούλους αρκετά ε, νωρίς ώστε να έχετε ήδη αποφανθεί. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο γιατί ε, κάνετε τις καταληκτικές παρατηρήσεις σας ως εισηγητής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Την κυρία Κλεβακέκους και τον κύριο Χρυσόγερο για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους που με ενισχύουν σε αυτά που και εγώ διαπίστωσα. Δηλαδή έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας, αλλά δεν αξιοποιούνται, διότι ο καθένας δουλεύει μόνο για την πάρτη του. Το παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχεδόν χωρίς επιτόκια, με ελάχιστο επιτόκιο, δίνει χρήματα στις τράπεζες και οι τράπεζες για λόγους των υποχρεώσεων σταθεροποίησης ε, και ρύθμισης που έχουν, τα κρατάνε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει εγγύησει που παρέχουν μακροπρόθεσμη ε, εγγύηση για ε, μεγάλων διαστάσεων προγράμματα. Και δεν αξιοποιούνται αυτές οι πιστώσεις. Γιατί δεν ξέρω. Μήπως δεν είναι γνωστές ή κάποιοι φοβούνται τους κινδύνους. Στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου αποφασίσαμε μια σαφή κατεύθυνση για αυτά τα διαθροτικά ταμεία. Θέλουμε βιώσιμη οικονομία, ενίσχυση μικρομεσαίων, ενίσχυση έρευνας και τεχνολογίας, διασφάλιση μεγάλων ε, ε, προγραμμάτων υποδομών κτλ. Οπότε θα έπρεπε αυτά τα όργανα, οι μηχανισμοί που έχουμε στη διάθεσή μας να βοηθήσουν τα κράτη που πλήττονται από την κρίση όπως το, ο μηχανισμός που αποφασίσαμε ε, για την κατανομή των κινδύνων που αφορούσε πολιτή προγράμματα. Δεν έχουμε πληροφόρηση για το τι έγινε με όλα αυτά τα μέσα, όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Γιατί είναι επαρκές πλαίσιο για να συνεχιστούν τα μακροπρόθεσμα μεγάλα προγράμματα. Αλλά αν αξιοποιούνται δεν το ξέρω. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι να υπάρχει μια συνολική επισκόπηση όλων των δυνατοτήτων και η βούληση και εδώ χρειάζεται δουλειά, η βούληση να, είναι πιο, ε, να ψάξει κανείς σε βάθος και να προσπαθήσει να προσαρμόσει τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση στις ανάγκες. Κάναμε ένα μεγάλο τμήμα, γιατί έχουμε τους νέους κανονισμούς για τα διαφθορτικά ταμεία Καθήκον λοιπόν τώρα της Επιτροπής μας, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι, είναι τώρα, τα επόμενα χρόνια, να ελέγξουμε οι δυνατότητες που δίνουν η Ευρωπαϊκή Θεσμική Ένωση πώς θα αξιοποιηθούν από τα κράτη-μέλη και κυρίως πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προωθήσουν αυτές τις δυνατότητες στις περιφέρειες, στις επιχειρήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 είναι η ημερομηνία και ψηφίζουμε στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Πάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. 7η και 8η έκθεση προόδου σχετικά με την πολιτική συνοχής. Βίλια Σαβισάρ Τόμάστα. Είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ. Τη δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που θα βασιζόταν υποτίθεται αρχικά μόνο στην 7η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροποποιήθηκε όμως και αφορά και την 8η τελικά έκθεση πρόοδου, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, καθώς και τη Στρατηγική Έκθεση 2013 για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η πολιτική συνοχής είναι, έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνοχή, να μειώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ούτως ώστε για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι και να αξιοποιηθεί η επιτυχία των προγραμμάτων και των μέτρων, θα πρέπει να κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση που να βασίζεται σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία. Η οικονομική κρίση σταμάτησε τη διαδικασία συνοχής. Για να μην πω ότι την ανέτρεψε, την ανέστρεψε και έχει μεγαλώσει τις ανισορροπίες των περιφερειών. Έχουμε μεγάλες ανισότητες σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ. Μέχρι στιγμής η πολιτική συνοχής ε, καθόριζε κάποιους στόχους και θέλαμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Δίναμε μεγάλη έμφαση στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων των πόρων, αλλά δεν αξιολογούσαμε αρκετά τους στόχους. Η χρήση των ε, ταμείων φτάνει μέχρι το 50%. Η διαδικασία όμως είναι πολύ αργή. από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης μέχρι την παραλαβή των κονδυλίων και τη χρήση των κονδυλίων είναι απίστευτα μακριά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λαμβάνουμε τα κονδύλια της ε, συγχρηματοδότησης πιο γρήγορα. Τα προγράμματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ε, εξαρτώνται αποκλειστικά από τα ταμεία συνοχής και τα κονδύλια τους. Και επειδή δεν υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, υπάρχουν μόνο τα ταμεία συνοχής για χρηματοδότηση. Η στόχοι της στρατηγικής 2020 είναι πολύ σημαντική, αλλά μην ξεχνάμε και την ε, εδαφική, πολιτική και κοινωνική συνοχή και οικονομική φυσικά συνοχή. Τώρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε επενδυτικά προγράμματα στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια. Λόγω της κρίσης, ο αριθμός των κοινωνικά αποκλεισμένων αντόμων αυξήθηκε σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις, θα πρέπει να εστιάσουμε σε δικές πολιτικές που μας εξασφαλίζουν ευκαιρίες βιώσιμες και που εξασφαλίζουν βεβαίως την κοινωνική ένταξη. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε καλύτερα τα μέτρα και να τα συντονίσουμε καλύτερα. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες και εγώ στην έκθεση αυτή και βεβαίως θα περιμένω και τις ιδέες των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Τόμας Ντόιτς δεν είναι εδώ και δεν τον αντικαθιστά κανένας, άρα ο Γιάννης Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Για αυτή την έκθεση μιλάμε για ιστορικά πράγματα πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία που βλέπουμε στην 7η και 8η έκθεση προόδου. Εγώ νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε αυτά που ήδη έχει πει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την περίοδο 2014-2020 ανταυτού. Δηλαδή θα πρέπει να τονίσουμε τα σημεία που είναι σημαντικά για το μέλλον και να καθοδηγήσουμε τα στατιστικά στοιχεία τους ώστε να επιβεβαιώσουν αυτά που θέλουμε να πούμε. Ε, λέγονται κάποια πράγματα, αλλά η ευφυή εξειδίκευση, παραδείγματο χάρη, δεν αναφέρεται σε μεγάλο βάθμο. Θα έπρεπε να το τονίσουμε αυτό το ζήτημα. Το ίδιο για τις περιφερειακέ εταιρικέ σχέσεις, τι, ποια σημασία έχουν για το μέλλον. Ε, νομίζω κάποια τέτοια στοιχεία θα βελτιώσουν την έκθεση και θα πρέπει να διασυνδέσουμε αυτά που λέμε ε, μέσα στην έκθεση με αυτά που λέμε για την περίοδο 2014 ως 20, ούτως ώστε να ιεραρχήσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας για το μέλλον. Και ε, θα πρέπει να ε, στοιχειοθετήσουμε αυτά που λέμε ανατρέχοντας σε αυτή την 7η και 8η έκθεση. Αλλά μην ανησυχείτε, θα καταθέσω πιο συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ότζη. Ευχαριστώ. Ε, είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη η έκθεση προόδου και η έμφαση που δίνεται κυρίως στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Όπως είπαμε και επευκαιρίες προηγούμενης έκθεσης ε, του κυρίου ε, Γκοντμάνης. Αυτή η περίοδος ε, της πολιτικής ε, συνοχής ε, τι μας διδάσκει ότι οι αστικές και οι υπεραστικές περιοχές διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, θα έπρεπε στα πλαίσια της όλης διαδικασίας να εξετάσουμε εάν θα επηρεαστεί η χρηματοδότηση Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει ανεξαρτησία μέσα στο σύστημα, αν έχει κατοχυρωθεί, εάν έχουν ενταχθεί οι πολιτικές και στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές. Άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ΟΤΑ που ε, θα πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα για να υλοποιήσουν στρατηγικές και δεν πρέπει να βαρύνονται από επιπρόσθετο διοικητικό άχθος ε, λόγω της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων. Αυτά είχα να πω και χαίρομαι πάρα πολύ που εξετάζουμε αυτή την έκθεση. Θα υποβάλω τροπολογίες. Πρόεδρος, ε, δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Γουόλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το, την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε για αυτές τις τρεις εκθέσεις. Μία σύντομη παρατήρηση. Και οι τρεις εκθέσεις ε, είναι συναφείς, αλλά ασχολούνται με διαφορετικά στατιστικά στοιχεία. Για την 7η και 8η έκθεση πρόοδο εξετάζουμε στατιστικά στοιχεία ε, του, του ΑΕΠ και άλλα στοιχεία για την ανεργία, βασικά για, την, για κοινωνικά ζητήματα. Ε, και επί τη βάση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και όντως ε, και αυτό απηχεί τη συζήτηση για την προηγούμενη έκθεση του κ. Γκοντμάνης διαπιστώνουμε ότι οι επενδύσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε, υφίστανται πάρα πολύ μεγάλη πίεση μιλήσατε για τους συντελεστές συγχρηματοδότησης ήδη και νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις και της τωρινής προγραμματικής περίοδου η κατάσταση εξυπακούεται από την κρίση, από την κρίση ως προς τη δημόσια ε, χρηματοδότηση. Ε, τα εθνικά στατιστικά στοιχεία στη στρατηγική έκθεση που δημοσιεύσαμε τον Απρίλιο ασχολούνται με την εφαρμογή αυτή καθεαυτή των προγραμμάτων. Βασιζόμαστε στα στοιχεία για την εποπτεία, την παρακολούθηση δηλαδή της χρηματοδότησης, Πώ κινητοποιείται η χρηματοδότηση και ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα τη εφαρμογή τη πολιτική. Αυτή η δέσμη των εκθέσεων που έχετε λοιπόν ε, είναι, απαρτίζεται από συμπληρωματικές εκθέσεις, αλλά όχι υπανομοιότυπες εκθέσεις, είναι συμπληρωματικές. Αρχίζουμε να βλέπουμε λοιπόν κάποιες αποδείξεις για τις, τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθούμε. Βλέπουμε επίσης ότι η επιλογή των προγραμμάτων σε κάποια κράτη-μέλη ε, δεν ε, προχωρά όσο γρήγορα θα θέλαμε. Ε, επηρεάζεται από την κρίση, από την έλλειψη χρηματοδότησης και σε πολλές περιπτώσεις από την έλλειψη τοπικής ικανότητας να εκπονεί και να υλοποιεί προγράμματα. Βεβαίω είναι λένε της οικονομία, αλλά δεν είναι αυτό ο καταλητικός παράγοντας. Είναι η δυνατότητα εφαρμογής του συμβατικού δικαίου, παραδείγματος χάρη, σε τοπικό επίπεδο ή ε, ε, καθεστώτα για τις κρατικές ενισχύσεις ή συμμόρφωση με σχετικές υποχρεώσεις. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που τονίζουμε στρατηγική έκθεση είναι ότι η πολιτική που εφαρμόζουμε σχετίζεται με τον αναπρογματισμό, αναεπιμερισμό των κονδυλίων σε περιοχές που τα χρειάζονται για την τόνωση της αγοράς εργασίας, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων κτλ. Και όπως είπε η συγγήτρια, σχεδόν 50% των κονδυλίων δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμα, δεν έχουν απορροφηθεί, είναι στη διάθεση των κρατών μελών ε, κυρίως στις ε, περιοχές και τα κράτη-μέλη σύγκλησης. Αυτό που εκτιμήσαμε στη συζήτηση και το τονίζουμε και εμείς στην έκθεσή μας είναι ότι χρησιμοποιούμε και τη στατιστική τα στατιστικά στοιχεία τη 7 η και 8 η έκθεση, αλλά και τι πληροφορίε για την παρακολούθηση των τωρινών προγραμμάτων. Έτσι μόνο θα προετοιμάσουμε καλύτερα προγράμματα, καλύτερα στοχευμένα προγράμματα για το μέλλον και ε, ε θα πρέπει να ενισχύσουμε την αξιολόγηση των, των ε, προγραμμάτων που τρέχουν για να κατανοήσουμε πραγματικά τι λειτουργεί αισίω και υπό ποιε συνθήκε για να συνειδητοποιήσουμε και τι πρέπει να αλλάξει τελικά. Διαβλέπουμε πάντως ήδη τα ωφέλη αυτών των εκθέσεων προόδου και την ε, αύξηση της διαφάνειας ως προς την ε, εφαρμογή της πολιτικής. Να άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν 27 εθνικές εκθέσεις που είναι επίσης διαθέσιμες και επισέρχονται, ε, ξεπακούνται σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ανά κράτος μέλος και με χαρά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Επιτροπή σας και με στη διάθεσή σας αν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια, κυρία Ουσπάνοβα. Ε, Ευχαριστώ. Έχω άλλη μια ερώτηση για την Κομισιόν. Νομίζω ότι πολλά υπόθηκαν ήδη, ωστόσο στην πρόταση γνωμοδότηση που έχουμε ενώπιόν μας με ανησυχεί το σημείο 11 και 12 όπου αναφερόμαστε στην έλλειψη δεδομένων από την επιτήρηση αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική και από πολιτική άποψη, γιατί επίκυνται και οι ευρωεκλογέ. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή ξεκινάει και η επόμενη περίοδος προγραμματισμού των πολιετών προπτικών, θέλουμε να έχουμε σαφή αποτελέσματα και να εξαγάγουμε διδάγματα από το τι έγινε στην περίοδο που τώρα λύγει για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο εισηγητής. Είναι ανεπαρκή η συλλογή δεδομένων. Είχαμε ένα ανεξάρτητο πρόβλημα για τις στατιστικές. Έχουμε πει πως σημαντικές είναι στατιστικές. Οπότε, σύντομη ερώτηση προς την Επιτροπή. Τι δυνατότητες, τι εργαλεία έχετε για να έρθετε σε επαφή, κράτη, να έρθετε σε επαφή με τα κρατημένη. Για να μην έρχεστε εδώ να μα λέτε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, δεν έχουμε καλέ στατιστικέ. Για να βελτιώσουμε τι στατιστικέ. Να είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη περίοδο προγραμματισμού επιτέλους θα έχουμε το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας, θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε αυτή την ευελιξία όταν διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, ούτως ώστε να τις απαντήσουμε μαζί. Αυτή η παράγραφος, ειδικά η παράγραφος 11, κατά την άποψή μου, είναι υπερβολικά σκληρή. Όταν βλέπετε τον όγκο των στοιχείων που μπορέσαμε να ε, εξεργαστούμε ομαδικά ε, και που παρουσιάστηκαν, υπάρχει βεβαίως ε, περιθώριο βελτίωσης των στοιχείων που έχουμε λάβει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε τώρα και πιο πρόσφατα στοιχεία. Η στρατηγική έκθεση ε, βασίστηκε σε στοιχεία του 2011 και εκεί έχουμε ομαδοποιημένα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και έχουμε 400.000 θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν συνολικά. Ε, τα στοιχεία του 2012 μας δείχνουν ότι περίπου 580.000 θέσεις απασχόλησης έχουν δημιουργηθεί γενικά στην πολιτική και στα 27 κράτη-μέλη. Επομένως, τα στοιχεία βελτιώνονται ε, υπάρχουν βεβαίω αδυναμίε σε ειδικέ ε, περιοχέ, ειδικού τομεί, αλλά λαμβάνοντα υπόψη ότι τα δεδομένα για την παραγωγή αφορούν ε, την εθελοντική χρήση βασικών δικτών, σημειώνουμε πρόοδο. Και τελικά θα αποτελέσουν τη βάση της εξπός αξιολόγησης που αρχίζουμε να ετοιμάζουμε και πιστεύω ότι θα μας διδάξει πολλά σε διάφορους τομείς. Τη εκ των λοιπόν αξιολόγηση. Όταν κοιτάξτε, το πακέτο που σας παρουσιάσαμε, ε, είναι συμπληρωματικό. Ε, μιλάμε για μακροπεριφερειακές στατιστικές ε, και έχουμε και πληροφορίες σε ένα πρόγραμμα. Τώρα χρειαζόμαστε την αξιολόγηση, ούτω ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ των προγραμμάτων και, της, και την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών τάσεων. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό είναι ο στόχο τη εκ των υστέρων αξιολόγηση. Να συνδέσουμε δηλαδή τι ευρύτερε εξελίξει στην οικονομία στην, ε, και τι κοινωνίε με τι δραστηριότητε των προγραμμάτων. Φυσικά είναι σχέδιο κειμένου, γι' αυτό το σχολιάζω. Ορισμένα από τα στοιχεία είναι πιο αξιόπιστα από ότι υπενήσεται αυτή η παράγραφος. Έτσι. Ε, εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε να το συζητάμε. Μπορείτε να το σχολιάσετε, δεν είναι τελικό κείμενο, είναι σχέδιο κειμένου. Άλλα σχόλια παρακαλώ, αν όχι να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Για να μας απαντήσει την εισηγήτρια πιο σωστά. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και να κάνω κάποιες προτάσεις για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Αν κοιτάξετε την ε, επικεφαλίδα αυτής της έκθεσης, πρέπει να εστιαστούμε στην ε, ανάλυση που υπάρχει στην 7η και 8η έκθεση προόδου. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Περιμένω τις ε, προτάσεις σας και μπορούμε να τις προσθέσουμε προς την Επιτροπή και προς τον συνάδελφο Βλάσικ. Θα ήθελα να σας πω ότι για τη συλλογή των δεδομένων. Αν δεν συλλέξουμε δεδομένα, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν οι πολιτικές μας, οι πολιτικές μας και τις Κομισιόν τελικά επηρεάζουν κάτι. Έχουν κάποιο αντίκτυπο. Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις, ότι είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτήν την παράγραφο και ότι δεν έχουμε αρκετές στατιστικές, από τα έγγραφα της Κομισιόν και από τις εκθέσεις διαφαίνεται ότι δεν έχουμε τα δεδομένα, τέλος πάντων αρκετά συγκρίσιμα δεδομένα. Αυτό το σημείο, αυτό τονίζει, ότι χρειαζόμαστε συγκρίσιμα δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Και με βάση αυτά τα συγκρίσιμα δεδομένα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Στο μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να φτάνουμε σε κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αυτά από πλευρά μου. Περιμένω τι τροπολογίε σας και τη συζήτηση των τροπολογιών φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τον Ιανουάριο είμαστε πιο χαλαροί. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου ε, έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες. Μεσημέρι, έτσι. Θα σταματήσουμε τώρα την συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 με τους εθνικούς βουλευτές και με τον Επίτροπο Χάν για να συζητήσουμε τις προκλήσεις για την εφαρμογή ε, της πολιτικής και των μελλοντικών πολιτικών. Ευχαριστώ.